Okay. Λοιπόν, καλημέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Πρόκειται για μια έκτακτη συνάντηση. Πρέπει να εγκρίνουμε εκ νέου την ημερήσια διάταξη. Φαντάζομαι ότι την δέχεστε. Μια, δύο αναγγελίες του Πρόεδρου. Πρώτον, νέα προθεσμία τροπολογιών για το σχέδιο εκθέσεις για τα προγράμματα της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της ε, χρηματοοικονομικής έκθεσης και λογιστικού ελέγχου 2014-2020. Ο κύριος Στόλεγιαν, ηγητής, πρότεινε την, αναβο... την αναβολή της προθεσμίας. Η νέα προθεσμία είναι η 10η Ιουνίου 5 το απόγευμα. Θα σας στείλουμε και νέο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε ακόμα την άφηξη του κύριου Ασμούσεν. Θεωρήσω ωστόσο σκόπιμο να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του Επιτρόπου για να μην χάσουμε χρόνο. Ελπίζω ότι μέχρι να φτάσουμε σε ερωτήσεις θα έχει φτάσει και ο κύριος Ασμούσεν. Θα μου πούν σύντομα. Λοιπόν, καλωσορίζω τον Επίτροπο και τη απουσία του και τον κύριο Ασμούσεν στην Επιτροπή. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση τη με την Τρόικα, γιατί τα δύο τρίτα τη Τρόικα. Όπω προβλέπετε στο Τούπακ, παρότι προεξοφλούμε λίγο την ημερομηνία υλοποίηση τη συμφωνία αυτή. Θέλουμε να συζητήσουμε την Κύπρο σήμερα. Σε μελλοντικέ συναντήσεις με την Τρόικα θα μπούμε και σε άλλες συγκεκριμένες χώρες ή θα κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση. Πάντως θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες συναντήσεις για να δούμε καλύτερα τη διαδικασία και την μεθοδολογία που ακολουθείται εν γέννη και να είναι περισσότερο ενήμεροι οι πολίτες για το πώς γίνονται, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Με χαρά να σας αναφέρω ότι οι ερωτήσεις που ανήγγειλα χθε παρουσία του κ. Ντάισεμπλουμ που εστάλησαν σε όλους απαντήθηκαν από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας ε, στάλθηκαν χτες το βράδυ αργά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Ε, περιλαμβάνονται και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Περιμένω να μου δώσουν το ok για το καθεστώς του εγγράφου προς την ε, δημοσίευση στο ευρύ κοινό. Ως θα έρθει αυτό. Πρόκειται για μια κοινή απάντηση της Επιτροπής και της ΕΚΤ, παρότι κάποια θέματα όπως το ELA ε, απαντώνται στην πράξη μόνο από τον υπεύθυνο θεσμό. Σε ένα, ένας θεσμό, ένα θεσμικό όργανο. Όταν είναι ένα θεσμικό όργανο υπεύθυνο, η απάντηση είναι από αυτό το όργανο. Αλλιώ είναι κοινή. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω ότι απαντούν σε ορισμένα ερωτήματά μας. Το πιστεύαμε ότι θα έρθετε μέχρι το τέλος των ε, ανακοινώσεων του, της Προεδρού. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή ως ε, εκπροσώπου της Τρόικα και παρόντος στη συναντήση για την Κύπρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρεν και κατόπιν στον κύριο Ασμούσεν. Κατόπιν θα έχουμε πεντάλεπτες ερωταποκρίσεις με το νέο format. Δύο άτομα, ε, εάν ε, ζητάτε ε, θέλετε περισσότερα ερωτήματα και παίρνετε 4,5 λεπτά, πραγματικά δεν θα υπάρχει απάντηση. Καλό είναι να σας απαντηθεί η ερώτηση από αυτό που είναι κυρίως υπεύθυνο. Οι ερωταποκρίσεις λοιπόν θα είναι πέντε λεπτά. Εάν εσείς μιλάτε 4,5 η απάντηση θα κρατήσει μισό λεπτό. Και μπορεί να μην επιτρέψω να ξεπεραστεί πολύ ο χρόνος. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για την Κύπρο μας στείλατε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ε, στείλαμε απαντήσεις γραπτές ερωτήσεις αυτές, μπορείτε να τις συμβουλευτείτε. Αποφασίστηκε το πρόγραμμα αυτό και οθετήθηκε το Μάρτιο και περιμένουμε την πρώτη δόση στα μέσα Μαΐου, σε μερικές μέρες ουσιαστικά. Η δόση αυτή θα επιτρέψει στην Κύπρο να αποφύγει μια άτακτη χρεοκοπία, η οποία θα είχε δραματικές συνέπειες για τον κυπριακό λαό. Τα βασικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα. Για ποιο λόγο η Κύπρος βρέθηκε σε μια τόσο δεινή χρηματοπιστωτική κατάσταση, ώστε τελικά χρειάστηκε να ζητήσει ένα πρόγραμμα στήριξης και για ποιο λόγο χρειάστηκαν εννέα μήνες από το αίτημα το οποίο κατεβλήθη μέχρι να καταφύγουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το πρόγραμμα αυτό και ποια είναι τα βασικά στοιχεία του προγράμματος αυτού για τη χρηματοδοτική στήριξη της Κύπρου. Το βασικό γεγονός είναι ότι τα προβλήματα της Κύπρου συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών. Αρχικά είχαμε έναν υπερδιογκωμένο τραπεζικό τομέα, ο οποίος είχε πολλά κέρδη μέσω της προσέλκυσης ξένων καταθέσεων με πολύ ευνοϊκέ συνθήκες. Τα τραπεζικά προβλήματα επιδεινώθηκαν στη συνέχεια από ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου. Δεν υπήρχε επίση η απαραίτητη τραπεζική εποπτεία και επομένω οι μεγαλύτερε τράπεζε τη Κύπρου συσσόρευσαν υπερβολική έκθεση σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Κύπρο για τη συσσόρευση προβλημάτων ήδη πολύ νωρί. Στείλαμε προειδοποιήσει καθώ επίση και συγκεκριμένε συμβουλέ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραπεζικά προβλήματα καθώ επίση και οικονομικέ ανισορροπίε και όλα αυτά εμπεριέχονται στι συστάσει του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Ιούνιο του 2011. Όταν τον Νοέμβριο του 2011 ήρθαμε σε επαφή με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές λέγοντάς τους ότι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης θα ήταν τελικά αναπόφευκτο, θα ήταν μάλιστα αναπόφευκτο, εκτό και να αντιμετωπίσουν αμέσω τα οικονομικά αυτά προβλήματα που είχαν εσωρευτεί. Και τελικά η Κύπρος ζήτησε χρηματοδοτική στήριξη, αλλά τελικά μόνο τον Ιούνιο του 2012, πέρυσι δηλαδή. Είναι ατυχές το ότι χρειάστηκε πάνω από μισό έτος προκειμένου η Κύπρος να αποδεχθεί την δυνότητα τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς επίσης και την μη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Και είναι επίση ατυχές το ότι χρειάστηκαν άλλοι εννέα μήνες στην Κύπρο προκειμένου να καταλήξει μια συμφωνία με το Eurogroup. Να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ρόλο τη στα πλαίσια των προγραμμάτων ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα βασίζονται σε μια διακυβερνητική συνθήκη. Και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να λαμβάνει δράση εξ ονόματο των κρατών μελών τη Ευρωζώνη, ακόμα και όταν διαπραγματεύεται ένα μνημόνιο κατανόηση ω μέλο τη Τρόικα. Στόχο Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας της, προθε... και της συμφωνίας για το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Κύπρου έχει ουσιαστικά τρεις βασικές πτυχές. Πρώτον, θελήσαμε να βοηθήσουμε την Κύπρο να επιστρέψει στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεύτερον, να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα, τόσο στην Κύπρο βέβαια όσο και στην Ευρώπη. Και τρίτον, να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα του ευρώ καθώς επίση και τη ενία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σκληρά για μια πιο βαθμιαία προσαρμογή του κυπριακού τραπεζικού κλάδου και της πραγματικής οικονομίας της χώρας, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρέους, καθώς επίσης και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η αναποφασιστικότητα, οι καθυστερήσεις, αλλά και πολύ σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί, ουσιαστικά περιόρισαν πάρα πολύ τις εναλλακτικές λύσεις. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ήταν έτοιμα να χορηγήσουν χρηματοδοτική υποστήριξη της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κύπρος θα έπρεπε με τη σειρά της να κινητοποιήσει σημαντικούς εσωτερικούς πόρους προκειμένου να καλύψει το υπόλοιπο των χρηματοπιστωτικών της αναγκών μέσω δημοσιονομικών μέτρων και μέσω ενός επιμερισμού του βάρους με τους πιστωτές του τραπεζικού της τομέα. Το Μάρτιο η οικονομική κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που τελικά το σενάριο μιας πιο βαθμιαίας οικονομικής προσαρμογής δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί. Ιδίω η κατάσταση των τραπεζών επιδεινώθηκε σε καθημερινή βάση πάρα πολύ. Πολύ σύντομα λοιπόν έγινε σαφές ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου, η Λαϊκή, έπρεπε αμέσως να εξηγιανθεί. Ο κίνδυνος μιας ε, ολοκληρωτικής κατάρρευσης όλου τραπεζικού συστήματος της χώρας ήταν εμφανής, καθώς επίσης και εξαφάνιση καταθέσεων, καθώς επίσης υπήρχε ένας κίνδυνος ε, άτακτης χρεοκοπίας για τη χώρα. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα αποτελούσαν πραγματική καταστροφή τόσο για την Κύπρο και τον Κυπριακό λαό. Μια σημαντική απόφαση που λήφθη τη στιγμή εκείνη ήταν η περίφραξη, η οριοθέτηση μπορούμε να πούμε, των ελληνικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, πράγμα το οποίο ενθάρρυναν οι εταίροι της Τρόικα και το ότι εστέφθη με επιτυχία η δραστηριότητα αυτή ήταν καθοριστικό προκειμένου να εμφυσίσουμε νέα εμπιστοσύνη και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Τώρα εστιαζόμαστε περισσότερο στην εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας το οποίο πραγματικά θα υποστηρίξει την Κύπρο στο να διορθώσει τις υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μεταρρυθμιστεί ο τραπεζικός τομέας μέσω βαθιάς αναδιάρθρωσης, να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ε, το κατάλληλο υγιές επίπεδο των ε, δημοσίων οικονομικών και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την ε, οικονομική ανάκαμψη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε έναν μικρότερο αλλά πιο ανθεκτικό και πιο διαφανή τραπεζικό τομέα στη χώρα. Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος καθώς επίσης και η αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου αυτού αποτελεί σημαντικό στατικό στοιχείο, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον ESM. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται δίπλα στον Κυπριακό λαό προκειμένου να βοηθήσει στις δύσκολε αυτές στιγμές και προκειμένου να καταφέρουν να ανακτήσουν την οικονομία τους. Θα δώσουμε τεχνική υποστήριξη στην Κύπρο μέσω, ενός, μιας, μέσω μιας ομάδας υποστήριξης και βασιζόμαστε και στη δική σα υποστήριξη προκειμένου να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους για την Κύπρο πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, εν κατακλείδη, θα έλεγα ότι μπορούμε να αποκομίσουμε τουλάχιστον τέσσερα διδάγματα από την όλη κατάσταση. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τι εγγυημένε καταθέσεις. Ως προς αυτό, το Eurogroup και η Κύπρος έλαβαν γρήγορη διορθωτική δράση και τόνισαν ότι οι εγγυημένε καταθήσεις είναι όντω εξασφαλισμένες στην Ευρώπη. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια τραπεζική ένωση και όλα τα επιμέρου στοιχεία της όπως για παράδειγμα ένας κοινός μηχανισμός εποπτείας και ένας κοινός μηχανισμός εξυγίανσης, προκειμένου να καταφέρουμε να προλάβουμε στο μέλλον την ανάπτυξη τέτοιων μη βιώσιμων τραπεζικών τομέων όπως είδαμε στην Κύπρο, που έχουν βέβαια και πολύ αρνητικές συνέπειες για την κυπριακή οικονομία και να έχουν βέβαια κινδύνους και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εν γέννη στην Ευρωζώνη. Τρίτον, όταν πλέον είναι απόφευκτο και πραγματικά χρειάζεται μια χώρα χρηματοδοτική υποστήριξη, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνετε η απαραίτητη δράση το συντομότερο δυνατό. Όταν δηλαδή εντοπίζετε το πρόβλημα αυτό, όταν εντοπίζετε αυτή η ανάγκη, οποιοδήποτε καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και για την οικονομία και ιδιαίτερα επιζήμια για την κοινωνία. Τέταρτον, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα διαρθωτικά προβλήματα του συστήματος λήψης αποφάσεων όσον αφορά την ε, χρηματοπιστωτική βοήθεια, τη χορήγηση χρηματοπιστωτικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ιδιαίτερα. Χρειαζόμαστε μία ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θα πρέπει οι ε, νυν διακυβερνητικές διευθετήσεις να περάσουν πλέον στο κοινοτικό πλαίσιο και θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη λογοδοσία εμπλέκοντας περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να καταφέρουμε να ενισχύσουμε και την εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης, προκειμένου πραγματικά να μιλάμε και να είμαστε ενωμένοι σε διάφορα φόρα, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή το G20, όπου χρησιμοποιούμε κυρίως μέσα παγκόσμιας διακυβέρνησης στα φόρα αυτά. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια κάποια προσωπική τώρα παρατηρήση και να ολοκληρώσω κατά αυτόν τον τρόπο το λόγο μου. Για πέντε χρόνια εργάστηκα πολύ σκληρά ω επίτροπο για θέματα διεύρυνση και προσπάθησα να διευκολύνω την επανένωση τη Κύπρου. Λυπάμαι πραγματικά που δεν έχει επιτευχθεί κάποια αποφασιστική πρόοδος ακόμα. Σήμερα θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η επανένωση της νήσου θα έδινε μια πολύ ισχυρή όθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου. Πιστεύω ότι είναι τώρα πραγματικά η κατάλληλη στιγμή να δοθεί μια νέα πνοή στην διαδικασία εκείνη που θα οδηγήσει στην επανένωση της νήσου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Θυμόμαστε όσοι είμαστε εδώ τις προσπάθειές σας στην προηγούμενη θητεία της Επιτροπής. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας. Καλώς ήρθατε κύριε Σμούσεν. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την οικονομική βοήθεια στην Κύπρο. Νομίζω ότι ήδη ε, κάναμε κάτι παρόμοιο για την Ελλάδα. Τώρα είναι πιο συγκεκριμένη η βάση ε, που ε, θέτετε κι εσείς μετά το πακέτο το τούπακ, το διπλό ε, των δύο νομοθετημάτων. Η ουσία των συζητήσεων, η διαδικασία της λήψης αυτών των αποφάσεων συζητήθηκαν με, με έκφραση διαφορετικών απόψεων και εδώ. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την δυνατότητα να παρουσιάσω τις απόψεις της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚΤ και να συμμετάσχω σε δημόσια συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εταίρους από τη, της για την πολύ καλή συνεργασία. Ιδιαίτερα ευχαριστώ προσωπικά τον Όλη Ρεν και την ομάδα του για τη δουλειά που κάναμε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πριν ε, συζητήσουμε για τα βασικά στοιχεία του προγράμματος προσαρμογής, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς η Κύπρος έφτασε καταρχήν σε μια τόσο δύσκολη θέση. Γιατί ανισορροπίες τέτοιας τάξης μεγέθους ε, αναπτύχθηκαν, γιατί τις άφησαν να αναπτυχθούν και ποια, γιατί είναι τόσο εξαιρετικής φύσης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Είναι ουσιώδεις αυτές οι ερωτήσεις και ελπίζω να τις ε, συζητήσουμε σήμερα και μετά τις ε, πρώτες παρατηρήσεις του Επιτρόπου Ρεν, εγώ θα επικεντρωθώ στον τραπεζικό τομέα. Στη δεκαετία του 2000 η κυπριακή οικονομία εξελίχθηκε προς ένα ε, μη ισορροπημένο επιχειρηματικό μοντέλο με υπέρμετρο βάρος στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η χώρα στόχευε να γίνει από τις πρώτες στην παροχή διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών. Οι κυπριακές τράπεζες προσήλκησαν μεγάλες εισρωές ξένων καταθέσεων ε, δραματικά επέκτηναν τους ισολογισμούς τους τα τελευταία χρόνια και ε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το συνολικό τραπεζικό σύστημα εκπροσωπούσε πάνω από το 700% του ΑΕΠ και σε σχέση με την απασχόληση κάθε τρίτη θέση εργασίας ε, αφορούσε τον χρηματοοικονομικό και τον τριτογενή τομέα. Μια ενεργός χρήση των σχετικών και σημαντικών εργαλείων της πολιτικής θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει μπορέσει να περιορίσει αυτές τις μη βιώσιμες εξελίξεις. Η προληπτική εποπτεία όμως ήταν πολύ αδύναμη και δεν εμπόδισε την συσσόρευση μεγάλων ανισορροπιών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η αύξηση του ενεργητικού ξεπέρασε τις εισρωές ε, των καταθέσεων και έτσι όλο και περισσότερο οι τράπεζες έγιναν ευάλωτες σε σχέση με τη χρηματοδότησή τους. Προσπάθησαν να προσελκύσουν ε, με καταθέσεις με υψηλά επιτόκια, κατά μέσον όρο κατά 2% υψηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Η εγχώρια επέκταση των πιστώσεων και οι μη σόφρονες πρακτικές δανειοδότησης πυροδότησαν μια φούσκα ακινήτων στην Κύπρο και όταν έσπασε η φούσκα αυξήθηκαν δραματικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επίσης οι κυπριακές τράπεζες ε, υπέστησαν μεγάλες ε, ε, απώλειες μετά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και αυτό επιδίνωσε ακόμα περισσότερο την κατάσταση των ισολογισμών. Η στρεβλή φύση του οικονομικού μοντέλου δεν περιορίστηκε στο τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, ε, σημαντικές εξωτερικές και εσωτερικές ε, ανισορροπίες ισορρεύθηκαν, όπως είπε και ο Επίτροπος Ρέν πριν από λίγο, δηλαδή ε, επίμονα ελλείμματα τροχούσων συναλλαγών, σημαντικές απόλυτες στην ανταγωνιστικότητα, αυξανόμενα δημόσια ελλείμματα, δημόσιο χρέος. Όλα αυτά άφησαν την Κύπρο σε αδύναμη θέση και δεν μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τραπεζικού της τομέα. Και αυτά τα προβλήματα φάνηκαν να είναι δραματικά, ιδιαίτερα συγκρινόμενα με το μικρό μέγεθος της οικονομίας. Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες που ε, καλύπτουν το μισό από τον ε, ε, εθνικό τραπεζικό τομέα είχαν εξελικτικά κεφαλαιακές ανάγκες περίπου 8 δις, δηλαδή περίπου το 44% του ΑΕΠ. Και αυτό έδειξε το Φεβρουάριο του 2013 η ανεξάρτητη διαδικασία δέουσας επιμέλειας. Αν το δημόσιο, αν το κράτος ε, είχε υπομειστεί αυτές τις μεγάλες ανάγκες ανακεφαλαιοποίηση, το χρέος θα είχε ανέλθει στο 145% του ΑΕΠ. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Παράλληλα, οι παραδοσιακοί τρόποι επιμερισμού του βάρους από ε, τους επιστοτές του ε, τραπεζικού τομέα, του, τους ιδιώτες επιστοτές, ε, θα ήταν περιορισμένες. Όλα αυτά έκαναν πάρα πολύ μεγάλη την πρόκληση και Τη κατάσταση τη Κύπρου, μια εξαιρετική κατάσταση, πρέπει να έχουμε υπόψη μα τις αρχικές συνθήκες όταν μιλάμε για το σχεδιασμό του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, αυτά θα αναφέρω τώρα. Ε, Τρει βασικοί στόχοι καθόρισαν τι διαπραγματεύσει για το μνημόνιο. Πρώτον, θα έπρεπε να μειωθούν οι κίνδυνοι από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεύτερον, θα έπρεπε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέου. Και τρίτον, να αποκατασταθούν οι συνθήκε για βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Συνδυάζοντα αυτού του τρει στόχου, ε, ε, ο συνδυασμό αυτών των τριών στόχων απεδείχθη μεγάλη πρόκληση για να το πω ήπια. Όχι μόνο το πρόγραμμα έπρεπε να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ε, βραχυπρόθεσμες ε, ανησυχίες σχετικά με την ε, δημοσιονομική σταθερότητα και την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αλλά έπρεπε να τοποθετηθεί σε πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να τύχει της ομόφωνης απόφασης από την Ευρωζώνη και τους μηχανισμούς του ESM. Η... Λόγω των εξαιρετικών οικονομικών και πολιτικών συνθήκων, διαπραγματεύσει τράβηξαν πολύ και έγινε κρίσιμη η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα. Έπρεπε η ΕΚ να αναλάβει δράση. Ο, Ο ΕΛΑ σκοπό έχει ε, να ε, στηρίξει ε, στα προβλήματα ρευστότητα στις ε, αξιόπιστης φερέγγιες τράπεζες χωρίς προοπτική ανακεφαλαιοποίηση, οι δύο μεγαλύτερε και πιο αδύναμες κυπριακές τράπεζες δεν θα μπορούσαν πια να θεωρηθούν φερέγγιε αξιόχρεε. Επίσης, ε, ε, η παροχή έλα σε αυτές τις τράπεζες δεν θα ευθυγραμμιζόταν με τους κανόνες του ε, συστήματος της Ευρωζώνης και, με τις διατάξεις της συνθήκη. Έτσι, η έκτα αποφάσισε στι 21 Μαρτίου ότι ο έλα θα συνεχιζόταν μόνο και μόνο εάν υπήρχε πρόγραμμα το οποίο θα διασφάλιζε ε, την φερεγγιότητα των σχετικών των συγκεκριμένων τραπεζών. Μετά τη συμφωνία του Eurogroup 25 Μαρτίου, η ΕΚΤ δεν έφερε αντιρρήσεις στο αίτημα για παροχή ΕΛΑ, δηλαδή ε, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στις δύο περιπτώσεις η ΕΚΤ έδρασε αυστηρά ευθυγραμμιζόμενη με τον κανονισμό της ε, εφήρμοσε τους υφιστάμενους κανόνες. Τίποτα περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Και τέλος, το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε ευρωπαϊκή Ένωση ε, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αντικατοπτρίζει, αντανακλά τους τρεις στόχους που προανέφερα. Ειδικότερα αποφασίστηκε να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των δύο μεγαλύτερων τραπεζών αποκλειστικά με ε, συμμετοχή των μη ασφαλισμένων ε, καταθετών και των... Ε, ε, θα έπρεπε να μην ε, βρεθούν οι πιστωτές των δύο τραπεζών σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι σε περίπτωση ρευστοποίησης. Θα έπρεπε επίσης, αυτό ε, είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Επίσης, ε, θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των συνθήκων για βιώσιμη ανάπτυξη, ισορροπημένη ε, ανάπτυξη. Από το 550 θα έπρεπε να περιοριστεί ο τραπεζικός τομέα στο 350% του ΑΕΠ στην αρχή του προγράμματος. Αυτό ε, είναι απαραίτητο για να ε, μειωθούν ε, οι υποχρεώσεις από τις τράπεζες προς το κράτος. Το πρόγραμμα επίσης προβλέπει πλήρη προστασία των καταθέσεων κάτω από 100.000 ευρώ που δεν θα υφίστανται απώλειες από τη στρατηγική της εξυγίανσης. Παρά τα πρωτόγνωρα μέτρα που ελήφθησαν μέχρι τώρα, το τραπεζικό τομέα ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η ρύθμιση επιμερισμού του βάρους επηρέασε αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταθετών και απέτησε την εφαρμογή προσωρινών και αναλογικών ε, κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στις αναλήψεις των καταθέσεων. Η βραχυπρόθεσμη κίνδυνη είναι υψηλή, επειδή η βαθιά ύφεση αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τους ισολογισμούς των τραπεζών η, ε, η στήριξη της μεγαλύτερης τράπεζας στον ΕΛΑ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Έτσι χρειάζονται σταθερά βήματα για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ε, χρηματοπιστωτικού τομέα και να ε, επαναοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη ε, στη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία της Κύπρου. Και νομίζω ότι η περίπτωση της Κύπρου ε, θύμισε σαφώς πόση σημασία έχει να έχουμε ε, ε, θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης του ταχύτερο δυνατόν γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σπάσουμε την αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίου και των τραπεζικών συστημάτων. Καταρχήν κατεδείχθη ότι η ταχεία ε, θέση σε ισχύ και εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού του SSM είναι σημαντική. Η συγκεντροποίηση της ε, ε, εποπτείας, όπως και η αποτελεσματική χρήση των προληπτικών, μακροπροληπτικών μέτρων, θα βοηθήσει να, και θα προλάβει την συσσόρευση ανισορροπιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα από νωρίς. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έναν ισχυρότερο, ε, βιωσιμότερο ε, τομέα χρηματοπιστωτικό που θα μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερον, κατεδείχθη ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντω ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εξυγένση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή ε, σειρά ε, κοινών ε, εξάντε κανόνων για το bail-in, για bail-enable περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία του ενεργητικού και προτίμηση καταθετών. Σε σχέση με το τελευταίο, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να θέτει τους καταθέτες στην κορυφή της ιεραρχίας των πιστωτών και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ρόλος του DGS στην εξυγένση θα περιορίζεται στην διασφάλιση των ε, καταθετών, ε, των επιλέξιμων καταθετών. Αυτό θα συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ε, με νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα στην εξυγίανση. Ε, περνώ έτσι στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης που είναι σημαντικός πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης και ε, συμπλήρωμα στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Απαιτεί ισχυρή ε, ε, αρμοδιότητα ε, και εξουσία στο επίκεντρό του που θα ελαχιστοποιεί το κόστος της εξυγίανσης και θα προβλέπει αμερόληπτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγίανσης το οποίο θα έχει πρόσβαση σε ε, στήριξη προσωρινή και δημοσιο... Ε, ε, ουδέτερη από άποψη προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στην πρώτη ερώτηση. Ο κ. Ζαν για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προς τον κύριο Ρέν απευθύνομαι αρχικά. Πρώτον, για να του πω ότι εκτίμησα τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε την κατάσταση. Μπορώ κάλλιστα να υποστηρίξω τα διδάγματα που αντλεί από την κρίση και τις ε, προβλέψεις που κάνει παρόμοιες με αυτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άλλωστε. Η μόνη μου ερώτη, το μόνο μου ερωτηματικό είναι αν η Κομισιόν θα έχει τη βούληση και τα μέσα να παροτρύνει, να οδηγήσει τις κυβερνήσεις να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα αυτό που μπλοκάρει την Ευρώπη σήμερα είναι οι θέσεις των κυβερνήσεων, των κυβερνώντων των οποίων και όπου βλέπουμε τα όρια της διακυβερνητικότητας. Μια παρατήρηση στο περιθώριο της Κύπρου. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι δεν, δεν είχε προβλεφθεί και μετρηθεί επαρκώς ε, το τι θα γινόταν. Οι συνέπειες του τι θα γινόταν η ότι η Κύπρος απέκρυψε την, την πραγματική κατάσταση, κάτι που οδήγησε σε καθυστερήσεις με δεδομένη την επικαιρότητα θέλω να σας προειδοποιήσω κατά του τρόπου που ερμηνεύονται ορισμένε αποφάσει επιτροπή σε κάποιε χώρε, μεταξύ των οποίων μία που γνωρίζω πολύ καλά, Ιδίω ό,τι αφορά τι προθεσμίε που, απε, που δίνονται σε κράτη για να αποκαταστήσουν τα οικονομικά του. Έχω την εντύπωση ότι αν η Επιτροπή έδωσε προθεσμία για αποκατάσταση τη οικονομική σταθερότητα ήταν για να επιτραπεί μια αποτελεσματική προσγείωση σε εύλογο χρόνο και για να τηρηθεί ο προβλεπόμενο στόχο. Η χρήση ωστόσο κάποιων φράσεων του Προέδρου Μπαρόζο και το ιδιαίτερο κλίμα για την Γαλλία στην Γαλλία για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα σημαίνει σήμερα ότι παρουσιάζεται η επιμήκυνση της προθεσμίας ως μια βασική αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής ότι αφορά την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Δεν σας ζητώ να λάβετε θέση επ' αυτού. Σας λέω να ζητήσετε από τους υφιστάμενους τους ή τους υπαλλήλους που βρίσκονται στις ενδιαφερόμενες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μια ε, πολύ καλή αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, να μάθετε τι γίνεται εκεί και να ενημερώνεστε πολύ ξεκάθαρα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής ούτω ώστε να μην ε, οδηγηθούμε με υποκρυπτόμενο τρόπο σε προβλήματα ερμηνείας που αφορούν και τις ενδιαφέρομενες χώρες και την Ευρωζώνη. Αν η Επιτροπή εφαρμόσει τα διδάγματα που αντλεί με διάβια, νομίζω στο κοινοβούλιο, του στην ομάδα μας, θα βρείτε την βασική, ε, την αναγκαία υποστήριξη. Ευχαριστώ. Δεν υπήρχε ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε πάντως, κύριε Ρέν. Κάνα δύο ερωτήσεις τις, διέβλεψα και ευχαριστώ για το σχόλιο και τις πληροφορίες που μου δίνετε. Η απάντησή μου αν η Επιτροπή έχει, στο ερώτημα αν η Επιτροπή έχει τη βούληση και τους πόρους να επηρεάσει τα κράτη-μέλη, είναι, έχει ως εξής. Βούληση, ναι. Πόρους, ε, κάπως. Και το εξηγώ. Δίνοντάς σας το ιστορικό της δημιουργίας του μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η κρίσιμη απόφαση λήφθηκε το Μάιο του 12, του 10, συγγνώμη. Η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού δημοσιονομικής σταθερότητας βάσει ενός προπολογισμού της Ένωσης και με μια σειρά πέραν αυτού σημαντικών εγγύσεων που θα είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο, σε κοινοτικό πλαίσιο. Την νύχτα της 9 προς 10η Μαΐου και το πρωί της μέσης εκείνης η κατάσταση είχε αλλάξει. Είχαμε το EFSM που είναι κοινοτικό εργαλείο με 60 δις και το EFSF που είναι διακυβερνητική ρύθμιση με 440 δισεκατομμύρια. Και δυστυχώς το EFSF δεν ήταν τόσο ισχυρό και ως προς τις αποφάσεις και ως προς τους πόρους που θα ήθελε η Ευρωζώνη για να, για να αποκαταστήσει την ε, δημοσιονομική σταθερότητα σε μόνιμη βάση. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την αρχική απόφαση. Εμείς δουλεύουμε σε αυτό το πλαίσιο. Και όπως εξήγησα, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής βοήθειας η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος όλων των κρατών μελών. Um, Ευχαριστώ η Ελίσσα Φερέιρα από τους, ε, από τους Σοσιαδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα της Κύπρου μας υποχρεώνει να αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα τρέναρε για 1,5 χρόνο και κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής ξεκινήσαμε μια σειρά νέων προτάσεων για την Τραπεζική Ένωση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πώς εξηγείται το ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος τη στιγμή της αλήθειας όμως υπήρξε τόσο λίγος συντονισμός και λήφθηκαν αποφάσεις που αμφισβήτησαν, που έθεσαν επαμφιβόλο ό, όσα ξέρουμε για την ανάγκη διαχωρισμού ε, τραπεζών κρατών και προστασίας των καταθέσεων και κάτω από 100.000 ευρώ. Η ιεραρχία της τράπεζας και οι μέτοχοι είχαμε πει ότι θα πρέπει να είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι. Πώς υπήρξε τόσο μικρό συντονισμό δεδομένου του ότι κράτησε τόσο πολύ η συζήτηση. Δεύτερον, προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάνατε συστάσεις προς τα κράτη και τις τράπεζες ή ήταν συστάσεις που έγιναν μέσω των εποπτικών αρχών των, της, Εθνικής, της ε, Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, διότι οι τράπεζες ήταν στη βάση του προβλήματος. Ξέρουμε τι, τα stress test, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ρευστότητα των, ε, των τραπεζών στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατευθύνει τους τους οργανισμούς συστημικής ε, παρακολούθησης. Δεν θα έπρεπε να το γνωρίζει νωρίτερα, δεν θα έπρεπε να είχε επέμβει νωρίτερα. Προς τον ε, αντιπρόεδρο της Επιτροπής πρέπει να προστατεύσουμε το ευρώ. Δεν θα έπρεπε να προεξοφλήσουμε ε, το, τις επιπτώσεις της πρώτης απόφασης. Πώς λειτουργούν τα πράγματα στο εσωτερικό της Τρόικα. Αυτό είναι μια ακόμα ερώτηση. Συμφωνώ με τα διδάγματα που αντλήσετε πρέπει να αντικαταστήσουμε να, να αλλάξουμε τον τρόπο αποφάσεων της Τρόικα. Σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα προσαρμογής που είναι που, ανοίγει, που δίνει ένα άνοιγμα στα κράτη μέχρι και 15%. Χρειάζεται το 2 να αλλάξει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα που δεν θα να είναι δια, διακυβερνητικό αλλά σε ευρωπαϊκή ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πότε θα λήξει τελικά η ιστορία της Τρόικα. Ο κύριος Σασμούσεν πρώτος. Ευχαριστώ. For your question. Για την ερώτησή σας. Ρωτήσατε γιατί αργήσαμε τόσο και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο αναμεταξύ. Είπα ότι λόγω των εξαιρετικών πολιτικών και οικονομικών περιστάσεων στην Κύπρο αλλά και μέσα στην, ε, στο Eurogroup η διαπραγμάτευση των προγραμμάτων ε, καθυστέρησαν πάρα πολύ. Και εν τω μεταξύ η κατάσταση του τραπεζικού τομέα επιδεινώθηκε. οι κυπριακές αρχές είχαν ήδη ζητήσει τον Ιούνιο πέρυσι χρηματοοικονομική βοήθεια. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα μπόρεσε να κλείσει τελικά φέτος το Μάρτιο μόνο. Τούτο δεν ήταν δυνατό να γίνει, στο ένα μεταξύ δεν ήταν δυνατό να φτάσουμε σε μια συμφωνία μεταξύ Τρόικα και Κυπριακών Αρχών που να πήγαινε προς απόφαση κατόπιν στο Eurogroup δεν μπορέσαμε να συνάψουμε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης που θα μπορούσε να πετύχει τους στόχους που ήταν η περιστολή των κινδύνων και η αποκατάσταση βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν ήταν δυνατό. Όντως καθυστέρησε, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά δεν ήταν θέμα διαφωνιών μέσα στην Τρόικα που οδήγησε στην μακρά αυτή διαδικασία, αλλά ήταν υπερβολικά δύσκολο να συμφωνηθεί το πακέτο που θα καλύπτει όλους τους σημαντικούς στόχους με τις υφιστάμενες κυπριακές αρχές. Γι' αυτό καθυστέρησε τόσο το μνημόνιο συνεννόηση με το Eurogroup. Συμφωνώ ότι κράτησε πάρα πολύ και επιδίνωσε την κατάσταση του τραπεζικού τομέα. Στο αναμεταξύ, θέλω να διευκρινίσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δίνει συστάσεις στις ε, τράπεζες. Δεν είμαστε ακόμα εποπτεύουσα αρχή. Ένα από τα διδάγματα που ανέφερα είναι ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Διότι στην κατάσταση αυτή, στην περίπτωση αυτή, οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας τουλάχιστον θα βρίσκονταν υπό μία είναι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Και αυτό αποδεικνύει σαφώς τον επίγοντα χαρακτήρα να έχουμε έναν Ευρωπαίο επόπτη των τραπεζών. Μέχρι τώρα ο μηχανισμός, η εποπτεία γινόταν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Καταλαβαίνω το ερώτημά σας πότε θα τελειώσει η Τρόικα. Και όλοι το τόνισε και σωστά ότι αυτό θα ξεκινήσει όταν το ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, γίνει απλήρως ευρωπαϊκός θεσμός. Είναι διακυβερνητικό εργαλείο που δημιουργήθηκε γιατί δεν είχαμε άλλο εργαλείο διαχείρισης κινδύνων. Έπρεπε να γίνει γρήγορα στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθήκων και εγώ δεν κατακρίνω το ESM. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Δεν υπήρχε αυτό το εργαλείο πλήρων. Ωστόσο, η διάρθρωσή του είναι κάτι αλόκοτο που δημιουργήθηκε για την ανάγκη διαχείρισης κινδύνου. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι τώρα αυτό το εργαλείο μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν θα πρότεινα να αλλάξουμε τώρα το σύστημα της Τρόικα μεσούσης της κρίσεως. Διότι παρότι ακούμε διάφορα αναπεριπτώσεις, κατά την άποψή μου και είχα εμπλακεί σε πολλές τέτοιες συζητήσεις Τρόικα, η Τρόικα έχει δουλέψει αρκετά καλά. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπετε διαφορές μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων, αλλά το βλέπεις και στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Είναι λογικό. Άλλοι να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην χρηματοοικονομική σταθερότητα, άλλοι στην, μεγαλύτερη, στην αύξηση της ανάπτυξης. Το βλέπεις αυτό και στο εσωτερικό του, του Δέλτα Νιτάφ σήμερα. Δεν θα άλλαζε λοιπόν την Τρόικα στο μεσούση τη κρίση, διότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση σήμερα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θα συμφωνούσα μαζί σα ότι πρέπει να επανέλθουμε σε μια πλήρως ευρω... σε ένα πλήρως ευρωπαϊκό σύστημα που να περιλαμβάνει και λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που θα θέτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κέντρο των δράσεων. Όλοι θέλεις και εσύ να πεις κάτι. Γιατί απαντήθηκε η πτυχή της ερώτησης που είχε να κάνει με την Τρόικα. Μα συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γιώργο. Και ουσιαστικά να απαντήσω περισσότερο στην ερώτηση της κυρίας Φερέιρα για ποιο λόγο χρειάστηκε τόσος χρόνος. Ο Γιώργο έχει δίκιο. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την κατάσταση στην Κύπρο, όσο και με την κατάσταση στην Ευρωζώνη. Στην Κύπρο και μιλάω έχοντας κάποια πείρα όλα αυτά τα χρόνια στην διαχείριση του κινδύνου είδαμε ότι ουσιαστικά είχαμε μια χώρα, τη συνήθι περίπτωση μιας χώρας που βρίσκεται μπροστά σε μια ανυπέβρελτη δεινή οικονομική κατάσταση που οδηγεί σε πρόγραμμα στηριξη τελικά. Καταρχάς, υπήρχε μια στάση άρνησης της πραγματικότητας, του μεγέθους του προβλήματος και αυτό από μόνο του οδήγησε καθυστερησει και στη συνέχεια άρχισαν να διαραίουν διάφορες χρηματοδοτήσεις από τη χώρα και το 2011 η Κύπρος κατάφερε τελικά να έχει ένα δάνειο από τη Ρωσία, κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο χρόνο, αλλά δεν χρησιμοποίησε το δάνειο αυτό και το χρόνο αυτό προκειμένου να καταφέρει να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα, δηλαδή τις μεγάλες οικονομικές ανισότητες που υπήρχαν στη χώρα. Και στη συνέχεια οδηγηθήκαμε στις διαπραγματεύσεις αλλά με πολύ πιο περιορισμένες προοπτικές πια. Νομίζω λοιπόν ότι η δέσμη των δύο μέτρων, το, δύο, το θα μας δώσει περισσότερες δυνατότητες και με μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Τώρα, συμφωνώ ότι προφανώς θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της ε, Ευρωζώνης. Η όλη διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη και για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όχι μόνο στα εθνικά τους κοινοβούλια, τα οποία θέσανε πολύ αυστηρές απαιτήσεις για το όλο πακέτο, αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που μιλάμε για την αναδιάρθρωση της Οικονομικής και της Νομισματικής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες λήψης αποφάσεων για την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταφέρνει με ειδική πλειοψηφία να λαμβάνει αποφάσεις για χρηματοδοτική βοήθεια, για ποιο λόγο να μην κάνει κάτι τέτοιο και η ίδια η Ευρωζώνη από την απαιτείται απόλυτη ομοφωνία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να λειτουργούμε για την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στην Ευρωζώνη, αν μπορούσαμε να είχαμε για το ζήτημα αυτό ενισχυμένη πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία και όχι απόλυτη ομοφωνία. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις. Θα πρέπει να διευθετήσουμε όμως τώρα και το χρόνο ομιλίας που έχουμε μπροστά μας. Ενδεχομένως να μην καταφέρουν να δευτερολογήσουν οι ουσιαλιστές, για παράδειγμα, εξ ονόματος του, α, των φιλελευθέρων κύριος Σκυλακάκης έχει το λόγο. Thank you. And I would like to uh, thank both. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για την ειλικρίνεια των απαντήσεών τους. Βλέπουμε ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα επικοδομητικό διάλογο. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δύσκολη. Το ΕΛΑ δίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε προσωρινά σε τράπεζες οι οποίες προσωρινά δεν έχουν ε, ε, ρευστότητα, αλλά που είναι ε, φερέγγιες. Το ΕΛΑ ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικά προς τη λαϊκή. Χάρη όμως στην αγνώριση του πλήρου ποσού των ζημιών από το ελληνικό PSI, ο λόγος φερεγγιότητας της λαϊκή έπεσε κάτω από το κατόφλι το οποίο είχε θέσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στη συνέχεια αυξήθηκε το ΕΛΑ από 3,5 σε 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 3,5 σε 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ το μεγαλύτερο τμήμα αυτό το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012. Αυτό οδήγησε σε ένα ποσό που αντιστοιχούσε στο 50% στο ΑΕΠ της Κύπρου. Πότε ελήφθη ακριβώς η απόφαση για να αυξηθεί το έλα προς τη λαϊκή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βάσει ποιων κριτηρίων ελήφθη η απόφαση αυτή και βάσει ποιων κριτηρίων θεωρήθηκε εκείνη τη στιγμή ότι η λαϊκή ήταν εφερέγγια τράπεζα. Επίσης, εφόσον το συνολικό χρέος της Κύπρου και με το εφιστάμενο πρόγραμμα δεν επιτρέπει χρηματοδότηση του ποσού αυτού από το κυπριακό κράτος. Πώς επιτρέπεται το 50% του έπνιας χώρας να χρησιμοποιείται ως ιδιωτικός πόρος από μία τράπεζα για ένα ολόκληρο χρόνο. Συντοποιείται ουσιαστικά ότι με την με τον επιτρέπεται το 50% του ΑΕΠ να δυστυχεί ουσιαστικά σε έλα, σε μια αφαιρέγγια τράπεζα, να δίδονται σε μια αφαιρέγγια τράπεζα, αυξάνεται ακόμα περισσότερο εμέσως το χρέος μια χώρας χωρίς να υπάρχει έγκριση από το κοινοβούλιο της χώρας. Και καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα αυτά, τα 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ, πήγανε στον ιδιωτικό τομέα, σαν ανθρώπους ουσιαστικά πήραν αυτά τα χρήματα και φύγανε, αποχώρησαν. Νομίζω ότι αυτή είναι ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Σωστά είπατε ότι η πρόβλεψη του ΕΛΑ σκοπό έχει να στηρίξει φερέγγιες τράπεζες που προσωρινά αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Και είχαμε τρία διαδοχικά βήματα στην παροχή ΕΛΑ προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Το πρώτο βήμα το 2010 και το 2011 σταδιακά έχασε την πρόσβαση σε, δημόσι... σε ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης σε σχέση με την κρίση ε, χρέους στην Ευρωζώνη και απώλειες λόγω των ε, ελληνικών ομολόγων που είχε. Το Σεπτέμβριο του 2011 είχε πιο σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και ε, προβλήματα εγγυήσεων και ε, ζήτησε βοήθεια από την ε, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Το δεύτερο βήμα ήταν στο τέλος του 2011. Ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης των πλήρων απολειών από το ελληνικό PSI, και λόγω σημαντικής ε, αύξησης ε, των ε, δανείων ο δείκτης φερεγγιότητας της λαϊκής έπεσε κάτω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές ανάγκες που έχουν οριστεί. Στις 29 Ιουνίου του 2012 η, δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε ομόλογο για 1,8 δις νέων κεφαλαίων για την λαϊκή ώστε να αντιμετωπίσει ε, τις κεφαλαϊκές ανάγκες της. Στις 2 Ιουλίου του 2011 και εν ώψη ιδιαίτερα της μη χρηματοδοτούμενης φύσης αυτού του ομολόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΑ αποφάσισε να δώσει ε, να ε, αντιμετωπίσει την λαϊκή με βάση την αρχή της πρόληψης και προφύλαξης. Από τότε η χρηματοδότηση της Λαϊκής έγινε από τον ΕΛΑ ε, μέσω της ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας και ε, αντιμετώπισε τα προβλήματα λόγω της ε, ε, κροής των καταθέσεων. Οι κυπριακές τράπεζες που έπαιρναν έλα αργότερα αναγνωρίστηκε ότι δεν μπορούσαν να θεωρηθούν φερέγγι στα πλαίσια ενός προγράμματος για την Κύπρο γιατί δεν υπήρχε προοπτική αξιόπιστης ανακεφαλαιοποίησης χωρίς την ύπαρξη προγράμματος. Αυτό εξήγησα στην εισαγωγική μου παρουσίαση. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το Μάρτιο ε, στις 21 φέτος ε, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοίνωσε ότι η συνεχιζόμενη παροχή του ΕΛΑ θα μπορούσε να ε, γίνει μόνο αν υπήρχε πρόγραμμα για την Κύπρο, πρόγραμμα προσαρμογής που θα μπορούσε να, προβλέπει την ε, φερεγγιότητα των Κυπριακών Τραπεζών. Τι έγινε λοιπόν. Η εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων του ΕΛΑ, που είναι εθνικό καθήκον, ο ΕΛΑ, και η λογική που κατήσχησε δεν διέφερε από εκείνη που εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες. Η λογική εφαρμόστηκε με τον ίδιο τρόπο και στην ελληνική περίπτωση. Έλα, δίνει Κεντρική Τράπεζα μόνος όταν υπάρχει φερεγγιότητα ή όταν υπάρχει σαφής προοπτική ότι η συγκεκριμένη τράπεζα που παίρνει έλα μπορεί να ξαναγίνει φερέγγια η αξιόχρεη ε, ε, και ε, θα ανακεφαλαιοποιηθεί ως μέρος στα πλαίσια ενός προγράμματος προσαρμογής. Έτσι λοιπόν ήταν παρόμοια η κατάσταση στο βαθμό που η προοπτική υπάρχει για ανακεφαλαιοποίηση. Η Κεντρική Τράπεζα τότε μπορεί να παράσχει έλα. Αλλά, όπως ε, είπαμε και στα πλαίσια της ε, προηγούμενης ερώτησης, η διαπραγμάτευση του μνημονίου ε, κράτησε για πολύ μεγάλο διάστημα, υπερβολικά μεγάλο διάστημα και σε σχέση με άλλες χώρες. Και κάποια στιγμή δεν ήταν σαφές ότι ήταν ξεκάθαρη η προοπτική ύπαρξης προγράμματος ούτως ώστε να ξαναγίνουν ε, οι τράπεζες. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά δεν απαντήθηκε η ερώτησή μου. Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που έκανα. Είναι πολλές οι ερωτήσεις ε, που έχουμε. Θα πρέπει να επανέλθουμε ε, στην απάντηση γραπτός. Ναι. Κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Με κάθε σέβας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αγνοεί τις αλληλεο... αλληλεπιδράσεις και αμοιβέ διασυνδέσεις μεταξύ χωρών και τα ε, δημοσιονομικά θέματα. Γιατί αντιλαμβάνεται αυτές τις αλληλεπιδράσεις όταν είναι πολύ αργά. Την περασμένη εβδομάδα ε, ήταν προφανές ε, ότι οι κυπριακές ε, τράπεζες ήταν αφαιρέγγιες. Ε, όμως η ανακοίνωση γι' αυτό καθυστέρησε. Ε, ήδη είχαν χρησιμοποιηθεί κεφάλαια για το ελληνικό χρέος. Οι κυπριακές τράπεζες δεν είχαν εξωτερική στήριξη και το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης ήταν σαφές ότι θα έπεφτε βαριά στους ώμους του Κυπριακού κράτους. Επίσης, τρίτον, ήταν επίσης προφανές επειδή το μέγεθος του Κυπριακού τραπεζικού τομέα υπερβαίνει το εφταπλάσιο του ΑΕΠ, ήταν προφανές ότι το Κυπριακό κράτος δεν θα μπορούσε να αναλάβει από μόνο του την διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Όλα αυτά ήταν ξεκάθαρα πριν από πέντε χρόνια όμως δεν ήταν ξεκάθαρα από πέρσι, δεν ξεκαθάρισε η κατάσταση πριν από έξι μήνες. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η αλληλεπίδραση ε, μεταξύ ε, κρατών και τραπεζικών τομέων, ε, τομέα. Εσείς γιατί δεν το καταλάβατε από νωρίς. Και μια μικρή υποσημείωση, μια και έχω λίγο χρόνο. Η Σλοβενία που είναι το επόμενο θύμα τραπεζικής κρίσης Επί 22 χρόνια γνωρίζαμε ότι το Σλοβενικό κράτος δεν έκανε ποτέ σοβαρή προσπάθεια ανακεφαλοποίησης, καμία ιδιωτικοποίηση δεν έλαβε χώρα. Η εσωτερική διακυβέρνηση ε, είναι αδύναμη, δεν υπάρχει διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες και έχουν συσσωρεύσει τεράστιο ποσό, περίπου 25% του ΑΕΠ, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και εσείς ως Επίτροπος για τη Διεύρυνση τους βάλατε στην Ευρωζώνη και τους κάνατε δεκτούς σε αυτή τη λέσχη που τώρα ε, μολύνει τους υπόλοιπους. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις δεν ήταν ξεκάθαρες στο δικό σας το μυαλό από νωρίς. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν για τη Σλοβενία γιατί κάνατε πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και ένα πολύ αυστηρό σχόλιο. Η Σλοβενία έχει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, δηλαδή και προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και στα δημόσια οικονομικά. Τα εντοπίσαμε και τα υπογραμμίσαμε στην έκθεσή μας που υποβάλαμε στα πλαίσια των μακρο... της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες και περιμένουμε αυτές τις ημέρες αναθεωρημένο και πιστικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας από την Σλοβενία, το οποίο θα αξιολογήσουμε τις επόμενες εβδομάδες και θα επανέλθουμε στο τέλος του μήνα και στις 29 Μαΐου συγκεκριμένα όταν θα δημοσιεύσουμε τις συστάσεις για κάθε χώρα. Και τότε θα δούμε αν θα καταστούν αναγκαία περαιτέρω βήματα πάνω στη βάση του πόσο πιστικό, συγκεκριμένο και αξιόπιστο θα είναι το πρόγραμμα της Σλοβενίας για τις μεταρρυθμίσεις και τη σταθερότητα. Τώρα, για τη συσσόρευση μη βιώσιμων ανισορροπιών στην Κύπρο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ λυπηρό βέβαια ότι μας πήρε τόσο χρόνο μέχρι να κατανοήσουμε απόλυτα το γεγονός ότι η Κύπρος έχει ε, μεγάλες και μη βιώσιμες μακροοικονομικές ανισορροπίες στον τραπεζικό τομέα κυρίως. Και αυτό σχετίζεται εν με την φύση της τραπεζικής εποπτείας και του κανονισμού. Ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις ε, για μια μικρή χώρα ε, προκειμένου περί της εποπτείας του τραπεζικού τομέα που είχε αυτό το μέγεθος όπως αυτό στην Κύπρο που απαιτεί ιδιαίτερη επαγρύπνηση ούτω ώστε να αποφευθούν επενδυτικοί κίνδυνοι. Αυτό θα είναι και ζήτημα κέριο εις ό,τι αφορά το δημοσιονομικό σύστημα εποπτείας στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν για να αποφύγουμε και να προλάβουμε τη συσσόρευση τέτοιων ε, μη βιώσιμων τραπεζικών τομέων στο μέλλον χρειαζόμαστε την Τραπεζική Ένωση όπως επίσης και έναν αποτελεσματικό ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Προχωρούμε στους πρασίνους, ε, Φιλίπ Λάμπερτ. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε κυρία Μουσεν. Πρώτη φορά μπορώ να σας θέσω μια ερώτηση. Πρώτον, από την ΕΚΤ και όχι μόνο από την ΕΚΤ αλλά και από την μεγαλύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τη μεγαλύτερη ε, πιστοτική ικανότητα και όχι με την μεγαλύτερη όπως λένε πολλοί συμπατριώτες σας ε, οικονομική δύναμη. Μιλήσατε για τον τραπεζικό τον, ε, τομέα. Κατά την άποψή σας, ε, τι πρέπει να καταλήξω. Οι μικρές χώρε έχουν μικρές τράπεζες οι μεγάλες χώρε έχουν μεγάλες τράπεζες Αυτή είναι η λογική της εσωτερική αγορά. Τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η πρόβλεψή σα είναι να, ότι λέτε το ΑΕΠ της χώρας θα μειωθεί κατά 12,5% τα επόμενα δύο χρόνια. Εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο όταν το διαβάζω και έχω ένα πρόβλημα αξιοπιστία. Εδώ υπάρχει ένα μοντέλο. Στην Ελλάδα ήταν το ίδιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέμενε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν θα ε, χρεοκοπήσει, ενώ πολλοί έλεγαν ότι ναι. Και έχω το, ε, την εξή ερώτηση. Η, βιωσιμο, η ανάλυση βιωσιμότητας αν υλοποιηθεί από την Επιτροπή και καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μήπω γίνεται για να ταιριάζει σε ένα σκοπό και όχι για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, η, οικονομία, η οικονομία της Κύπρου πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα μειωθεί πολύ σημαντικότερα, ενώ η υποεκτίμηση της μείωσης κατά την άποψή μου φαίνεται να αιτιολογείται από το ότι δεν θέλουμε να καταβάλουμε την προσπάθεια στις πιστότερες χώρες τις μεγάλες πιστότερες χώρες. Το πρόβλημα όμως τόσο είναι ότι α, όταν τα σχέδια δεν είναι αξιόπιστα και δημιουργούν ε, στην αγορά και δεύτερον χρειάζεται να αναθεωρηθούν. Η ερώτησή μου είναι, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια, αυτή η κατάσταση άρνησης, ε, αυτή που χρησιμοποιεί και, και, και όλοι δεν, δεν είναι επι, ε, επιβαρυντικό όχι μόνο για τους λαούς της συγκεκριμένης χώρας αλλά και για όλες τις πιστότερες χώρες στην Ευρώπη. Mr. Lambert, thanks that you... Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ που ασκήσατε το προνόμιο να μου θέσετε για πρώτη φορά ερώτηση και για μένα είναι προνόμιο να σας απαντήσω για πρώτη φορά. Ναι, έχω γερμανικό διαβατήριο, αλλά η εντολή μου είναι ευρωπαϊκή και επ' αυτής ε, εδράζομαι. Για την παρατήρησή σας για το μέγεθος του τραπεζικού τομέα. είναι απλουστευτικό να κοιτάμε απλά μόνο το μέγεθος ε, του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ μιας χώρας. Αν ακολουθήσουμε την προσέγγιση αυτή, μπορούμε να συγκρίνουμε τη χώρα με, άλλες, ε, με άλλα υποτμήματα της νομισματικής ένωσης. Αυτή η προσέγγιση ωστόσο είναι απλουστευτική. Αυτό που έκανε εξαιρετική, μοναδική στην Κύπρο δεν ήταν μόνο το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, αλλά κυρίως η δομή των, του ενεργητικού και του παθητικού. Δηλαδή εμείς πρέπει να δούμε τα τροτά στοιχεία του τραπεζικού τομέα. Δεν ήταν ε, πρόθεσή μας να σταθούμε μόνο στην απλουστευτική προσέγγιση που προνέφερα. Θα συμφωνούσα μαζί σας ότι η άρνηση της πραγματικής κατάστασης πριν ή κατά τη διάρκεια ισχύω ενό προγράμματος, αυτό θα αυξήσει το κόστος για όλη την Ευρωζώνη. Όταν λοιπόν τέθηκε το ερώτημα στον όλοι σήμερα, γιατί η κατα τη διαρκεια ισχυω ενο προγραμματος αυτο θα αυξησει το κοστος για ολη την ευρωζωνη οταν λοιπον τεθηκε το ερωτημα στον ολη σημερα γιατι η επιτροπη δεν έκανε κάτι περισσότερο, την καθυστέρηση, ξέρετε καλύτερα από μένα τι έγινε στις διαπραγματεύσεις για το Τούπακ υπήρξε ένα σχέδιο προβλέψεων που θα έδινε την εξουσία στην Επιτροπή να πιέσει μια χώρα, να επιβάλλει σε μια χώρα ένα πρόγραμμα αν αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις υπόλοιπες ε, χώρες Ευρωζώνης. Αυτό το σχέδιο ωστόσο δεν επιβίωσε των διαπραγματεύσεων. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υποστηρίζαμε να είχε την εξουσία αυτή η Επιτροπή και το είπαμε στο Συμβούλιο αρκετές φορές. για τις παρατηρήσεις σας τώρα, ερωτήματα παρατηρήσεις ως προς τις ε, προβλέψεις για την ανάπτυξη της Κύπρου κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Είναι σωστό. Θα περιμέναμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα περισταλεί σημαντικά. Μείον 13% σωρευτικά για φέτος και του χρόνου ενώ η εσωτερική ζήτηση θα μειωθεί για την ίδια περίοδο, προβλέπεται να μειωθεί την ίδια, κατά 20%. Αυτή είναι κοινή προσθέση της πρόβλεψη της Επιτροπής και της ΕΚΤΟ ότι η οικονομία θα ανακάμψει το 2015 με δεδομένο ότι ένας μικρότερος και πιο ανθεκτικός τραπεζικός τομέα θα, θα αρχίσει να ξανά αναπτύσσεται. Είναι σαφές ωστόσο και είμαι ειλικρινής εδώ ότι και μέσο και βράχη και μέσο πρόθεσμα οι κίνδυνοι παραμένουν, υπάρχει κίνδυνος μείωσης ε, κάμψης οικονομικής που μπορεί να αντισταθεί, να, να ε, αλλάξει μόνο με ένα στέρεο πρόγραμμα εξυγίανσης. Υπάρχει και επιπλέον ε, αβεβαιότητα όταν κάνουμε τον υπολογισμό της μελλοντική οικονομικής ανάπτυξης, διότι αυτό που μπορούμε σίγουρα να αναμείνουμε είναι ότι η κυπριακή οικονομία θα πρέπει να μεταβάλει το επιχειρηματικό της μοντέλο, διότι το εφιστάμενο δεν ήταν βιώσιμο και αυτό το ζήτησαν πολλοί εμπλεκόμενοι. Να αλλάξει η χώρα το επιχειρηματικό της μοντέλο. Όταν αλλάζει ωστόσο το επιχειρηματικό μοντέλο αυτό απαιτεί διαρθρωτική τομή και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ενσωματώσει σε ένα εφιστάμενο οικονομικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν είναι και μια επιπλέον βεβαιότητα. Οι διαθροτικές αλλαγές στην οικονομία που καθιστούν δυσκολότερο. Δεν μπορείς να αλλάξεις μια οικονομία σε δύο χρόνια, αυτό θα ήθελα να σας πω. Περισσότερο χρόνο χρειάζεται. Ο κύριος Χουντής από την ΚΟΕ για την επόμενη ερώτηση. Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε να συζητάμε τώρα για την Κύπρο, τέταρτη χώρα υπό μνημονίου και υπό την εποπτεία της Τρόικα. Συζητάμε με τα δύο τρίτα της Τρόικα για την περίπτωση της Κύπρου. Δεν ξέρω ποια χώρα θα έχει σειρά, ήδη αναφέρθηκαν ορισμένες. Ο μηχανισμός στήριξης ο ευρωπαϊκός έγινε μόνιμος από το Σεπτέμβρη και διαθέτει δύο εργαλεία. Το ένα είναι δάνεια για τη στήριξη της σταθερότητας, σε χώρες που, δεν, που έχουν προβλήματα με τις δημοσιονομικές ανάγκες και ο δεύτερος δάνεια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στην περίπτωση της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι ε, υποδειγματικά θα έλεγε κανείς όσο αφορά τους δημοσιονομικούς δείκτες, ενδεχομένως καλύτερους και από τη Γερμανία, είναι το 16ο μέλος της Ευρωζώνης, επελέγει η τακτική του μνημονίου, το οποίο μνημόνιο και η τακτική της Τρόικα το οποίο ε, δένει χειροπόδαρα Κυπρίους και Κυπριακή οικονομία. Ξέρουμε την εμπειρία από τις χώρες που ήδη υφίστανται αυτές τις πολιτικές. Τώρα, τα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, αγαπητοί κύριοι, σχετικά με το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης για την Κύπρο. Μας έχετε μπερδέψει. Στην αρχή λέγαμε για 17,5 δις, αναφέρεστε τώρα, αναφέρετε για 23,5 δις. Πείτε μου τελικά πόσο είναι αυτό το ποσό, πώς το έχετε υπολογίσει. Από αυτό το ποσό ξέρουμε τα 10 πώς θα εξευρεθούν από, την Ευρωπαϊκή, από, τον, ε, από το Μηχανισμό Σταθερότητας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα υπόλοιπα 13 που πρέπει να προσφέρει η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία, ποιοι, από ποιους πόρους θα βγουν. Εδώ παρενθετικά, έστω και τώρα μπορεί η Κύπρος να διεκδικήσει αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων ύψους 4,5 δις. Και η δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Από αυτά τα 13 δισεκατομμύρια που ψάχνει σύμφωνα με τον προγραμματισμό σας να εξεύρει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι φανερό ότι θα υπάρξουν ιδιωτικοποίησεις στον ενεργητικό, στον, σε στοιχεία ενεργητικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το ερώτημά μου είναι αν σε αυτές τις ιδιωτικοποίησεις και θέλω να μου δώσετε σαφή απάντηση αν είναι δυνατόν περιλαμβάνονται και πιθανά μελλοντικά έσοδα της Κύπρου από την εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων όποτε και αν γίνει αυτή. Δηλαδή έχετε ζητήσει κάτι τέτοιο, θα το ζητήσετε ούτω ώστε να γίνει συνδιαχείριση αυτών των πόρων σε όφελος των δανειστών. Uh, Όλοι νομίζω ότι σε σένα απευθύνεται καταρχάς το ερώτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας κύριε Χουντή. Καταρχάς, αποφασίσατε, μας είπατε ότι αποφασίσετε να περάσουμε σε μνημόνιο. Είναι απόφαση της Κύπρου, είναι απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης αυτή. Εγώ θα προτιμούσα η Κύπρος να ήταν σε θέση να τα βγάλει πέρα με την οικονομική της κατάσταση χωρίς να καταφύγει σε κάποιο πρόγραμμα στήριξης. Αλλά αυτό δεν κρίθηκε δυνατό γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ ότι θα είχαμε μια άτακτη χροκοπία με δεινές συνέπειες για τον κυπριακό λαό. Όσον αφορά το ερώτημά σας για τις ανάγκες χρηματοδότησης, καθώς επίσης και για τους χρηματοδοτικούς πόρους, έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι ε, Υπάρχουν διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Αυτό οφείλεται όμω στο ότι καταρχά πολλοί συγκρίνουν διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Γιατί το πρώτο πρόγραμμα, και απλοποιώ κάπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή, και το κάνω αυτό για να σα εξηγήσω κάπω καλύτερα τα πράγματα. Η πρώτη απόφαση, που δεν ήταν βέβαια τελική απόφαση, ελήφθη πάνω σε καθαρούς όρους, ενώ η δεύτερη απόφαση περιείχε και ένα ποσό το οποίο δεν ήταν καθαρό, το οποίο ήταν μεικτό και είχε να κάνει με την κινητοποίηση εσωτερικών πόρων της Κύπρου όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης bail-in και εξυγίασης των τραπεζών της. Γι' αυτό το λόγο τα αριθμητικά δεδομένα παρουσιάστηκαν διαφορετικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Και ενώ αρχικά μιλούσαμε για 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους εσωτερικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού bail-in και της τραπεζικής εξυγίανσης, ουσιαστικά είχαμε θέσει έναν νότο ποσό 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού είχαν θέσει τα κοινοβούλια και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όσον αφορά την ερώτησή σας τώρα για τις ιδιωτικοποιήσεις και όσον αφορά τους υδραγανάνθρακες. Ως μέρος του προγράμματος αυτού κάποιες κρατικές επιχειρήσεις θα ιδιωτικοποιηθούν. Αυτό είναι μέρος της χρηματοδότησης του προγράμματος. Αυτό έχει αποφασιστεί και αποτελεί πλέον τμήμα του μνημονίου. Το ζήτημα τώρα των εσόδων από το φυσικό αέριο δεν θεωρούνται ως τμήμα του προγράμματος, αν αυτή είναι η ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Thank you. If we go on Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάγκεν εξ νόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την εντύπωση ότι η Τρόικα και όχι τα κράτη είναι υπεύθυνοι ε, για το τραπεζικό τομέα. Ε, αυτή είναι η εντύπωση που μου δώσατε. Η ευθύνη για την στρεβλή ανάπτυξη ε, αναλαμβάνεται από τα κράτη-μέλη. Και ο κύριος Ρένε είπε ότι πέρασαν 15 μήνες μέχρι να υπάρξει ανάληψη δράσης. Όπως και να το συζητάμε το θέμα, Ελίζα, η Τρόικα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η λύση. Όχι μόνιμη λύση, αλλά εκείνη πρόσφερε τις λύσεις. Αυτό το τονίζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις της Τρόικα θα πρέπει να ε, υιοθετηθούν χωρίς καμία κριτική. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Κομισιόν πρώτα. Πώς έγινε στο πρώτο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είχαν προταθεί να συμμετέχουν οι καταθέσεις από 25.000, ε, πράγμα το οποίο ε, κατέστρεψε την εμπιστοσύνη των καταθετών όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και δεύτερον, κύριε Άσμουσεν, δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο, φιλελε... ο συνάδελφος ε, από τους φιλελευθέρους ότι όσο διέθετε φθηνό χρήμα η ΕΚΤ, οι κυπριακές τράπεζες, ε, ε, τέσσερα δις τοξικά ομόλογα μπόρεσαν να αγοράσουν σε προβληματική φάση από την Ελλάδα. Δεν διέθεσε η ΕΚΤ αυτά τα χρήματα. Τώρα έχουμε την Κύπρο με 7 πλάσιο του ε, τραπεζικό τομέα, η Ιρλανδία με 12 πλάσιο, η Ιρλανδία τώρα είναι σε σωστό μονοπάτι, μειώνεται, θα μειωθεί ο τραπεζικός τομέας και στην Κύπρο. Στη Μάλτα 7 πλάσιο ο τραπεζικός, 27 φορές σε σχέση με το ΑΕΠ είναι ο τραπεζικός τομέας στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, Μπορείτε να μας δώσετε μια προοπτική κάτω από ποιες ε, συνθήκες είναι η ε, κατάσταση ε, επικίνδυνη όταν ξεπερνά τόσο πολύ ο τραπεζικός τομέας το ΑΕΠ και πότε μένει υπό έλεγχο. Όλοι να δώσω πρώτα σε σένα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συνεκτικός. Νομίζω ότι το βασικό το, ε, στην ευρύτερη εικόνα που παρουσίασε ο κύριος Λάνεν είναι ότι η μεταρρύθμιση της οικονομικής ε, διακυβέρνησης που κάναμε από κοινού και τη συνεχίζουμε από κοινού μέχρι τώρα εστιάζεται στην πρόληψη αυτών των οικονομικών ανισορροπιών που αποτελούν και το έναυσμα για την κρίση στην Κύπρο. Και η πρόληψη πάντα είναι καλύτερη από την διόρθωση όπως μάθαμε με σκληρό τρόπο. Και η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει την Ευρωζώνη να αποφεύγει τέτοιου είδους μεγάλες και μη βιώσιμες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τώρα, εις ό,τι αφορά το θέμα της λήψης αποφάσεων στην, ε, στο Eurogroup και αυτό ε, ήταν, αναφέρομαι στο πρώτο πακέτο που μετά τροποποιήθηκε με δεύτερη απόφαση. Όπως είπα, για διάφορους λόγους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας επί του Κυπριακού προγράμματος. Έγιναν πολλοί γύροι ε, συζητήσεων μεταξύ Τρόικα και Κύπρου σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη που όπως γνωρίζετε είναι οι ιδιοκτήτες του ε, ESM και που τον χρηματοδοτούν και που ορίζουν τις κρίσιμες παραμέτρους ε, ενό προγράμματος ε, χρηματοδότησης. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να πω ότι η αναποφασιστικότητα, οι καθυστερήσεις και οι μεγαλύτερες οι δημοσιονομικοί περιορισμοί επεριόρισαν τις επιλογές που ήταν διαθέσιμες κατά τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα κράτη της Ευρωζώνης ε, είχαν ε, αναφέρει βοήθεια 10 δις που ε, σήμαινε ότι θα, η Κύπρος θα έπρεπε να κινητοποιήσει σημαντικούς εσωτερικούς πόρους μέσα από μερικό στο τέλος η μη επίτευξη συμφωνίας θα ήταν χειρότερο πράγμα γιατί έτσι όλες οι καταθέσεις θα διέτρεχαν κίνδυνο στην Κύπρο εφόσον δεν θα υπήρχε ε, πρόγραμμα ε, προστασίας εγγύησης των καταθέσεων και θα ε, είχαμε οδηγηθεί σε χρεοκοπία του κράτους. Και αυτό θα ήταν χειρότερο και για την Κύπρο και για την Ευρωζώνη. Μετά την πρώτη απόφαση λοιπόν το Eurogroup ε, συνεδρίασε ε, πριν από την ψηφοφορία στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και σε αυτά τα πλαίσια η Τρόικα ομοφόνος, και το υπογραμμίζω αυτό, κατέστησε σαφές ότι εναλλακτική λύση χωρίς εισφορά στις καταθέσεις κάτω από τις 100.000 ευρώ ε, θα ήταν προτιμητέα ενώ θα σεβόμεθα τις ε, οικονομικές παραμέτρους που είχε θέσει το Eurogroup. Οι κυπριακές αρχές δεν δέχτηκαν αυτή τη σύσταση. Μετά χρειάστηκε ε, γρήγορη διορθωτική δράση από το Eurogroup και τις Κυπριακές Αρχές και όπως γνωρίζετε η τελική απόφαση δεν περιλαμβάνει την εισφορά αυτή και προστατεύει τις ε, επενδύσεις ε, όπως και πρέπει. Τις καταθέσεις, με συγχωρείτε. Ε, ο κύριος Άσμουσεν σε σχέση με την ρευστότητα, το Λουξεμβούργο, το Εύρος και το μέγεθος του τραπεζικού τομέα των χωρών. Ευχαριστώ κύριε Λάγεν για τις ερωτήσεις σας. Για το πρώτο μέρος σχετικά με την παροχή ΕΛΑ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ιδιαίτερα στη Λαϊκή, και το ερώτημα αν οι τράπεζες αγόρασαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό ε, ομολόγων όταν ήδη το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και οξύ. Ε, Έχω ήδη πει ότι ιδιαίτερα τη δεύτερη ερώτηση δεν μπορώ να την απαντήσω, γιατί ακόμα δεν έχουμε την θέση και το καθεστώς της εποπτικής αρχής. Δεν έχω λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με αυτό. αυτό που βλέπουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΕ ήταν ότι υπήρχε υποκεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αποκλείονταν από τις συνήθεις νομισματικές ε, ε, πράξεις και συναλλαγές και ε, έτσι πέρασε ε, ε, ε, πέρασαν στην παροχή του ΕΛΑ. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότης και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντιταχθεί με δύο τρίτα πλειοψηφία στην παροχή του ΕΛΑ μόνο αν η τελευταία δεν ευθυγραμμίζεται με, το, με τους συνολικούς στόχους της νομισματικής πολιτικής. Η εποπτεία της τράπεζας βρίσκεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τώρα για το ευρύτερο ερώτημα που θέτεται, τι κάνει έναν τραπεζικό τομέα ευάλωτο. Μη γελάσετε, θα το εξειδικεύσω αυτό λιγάκι, θα πω εξαρτάται. Δεν, δεν ε, είναι μόνο το μέγεθος του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ μιας χώρας που κάνει τη διαφορά ή δημιουργεί επικινδυνότητα. Αυτό είναι υπεραπλούστευση. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ο τραπεζικός τομέα στην Σλοβενία αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και χρειάζεται και θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα πρόσθετα κεφάλαια. Αλλά ο συνολικός τραπεζικός τομέας της χώρας είναι στο 150% του ΑΕΠ. Ενώ από την άλλη πλευρά απλά και το μέγεθος του τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ στην περίπτωση της Μάλτας, της Ιρλανδίας, και του Λουξεμβούργου ε, πραγματι έχει μέγεθος, αλλά δεν υπάρχει τραπεζικός τομέας στην ε, Ευρώπη που να ε, συγκρίνεται με το κυπριακό τομέα. Η Ιρλανδία, η Μάλτα, το Λουξεμβούργο δεν συγκρίνονται ε, ως προς τους τραπεζικούς τους τομείς με την Κύπρο, γιατί πρέπει να δούμε βαθύτερα την δομή τον του ενεργητικού και του, καθε, του παθητικού του τραπεζικού τομέα. Για να σας δώσω κάποια ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με το πώς η τροτότητα εξαρτάται. Εδώ πρόκειται για τομέα που προσελκύει πολλές ξένες καταθέσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη τροτότητας, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό όμως. Το θέμα είναι σε ποιο νόμισμα προσελκύεται καταθέσεις και σε ποιο νόμισμα ε, εκδίδεται τα δάνεια για να ε, εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για το συνολικό τραπεζικό τομέα. Επίσης πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα οι ισολογισμοί των τραπεζών επεκτείνονται, διογκώνονται. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα. Ε, πρόκειται για ρίσκο για τον εγχώριο, ε, τον εθνικό τραπεζικό τομέα ή ας πούμε είναι καλύτερη η κατάσταση στη Μάλτα όπου η πλειοψηφία των, του τραπεζικού τομέα είναι στα χέρια μεγάλων διεθνών τραπεζών που εσωτερικά μπορεί να προστατεύσουν καλύτερα εναντί κινδύνων τα υποκαταστήματα ή τις θηγατρικές τους σε μια χώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολλά επιμέρου στοιχεία τη δομή ενεργητικού και παθητικού και να μην περιοριστούμε μόνο στο συνολικό μέγεθο του τραπεζικού τομέα. Έχουμε πρόβλημα χρόνου, όπως βλέπετε. Δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ερωτήσεις, παρά μόνο εάν πιέσουμε λίγο το χρόνο. Ο κύριος Χάκμαρκ για το ΕΛΚ. Έφυγε. Η κυρία Κράτσα, θέλετε, εδώ έρχεται ο Γκούναρ, πού είναι. Uh, Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ήμουν έξω για άλλη δουλειά. Πρώτον, για το θέμα που μιλάμε, με την ευκαιρία θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί υπήρξε συμφωνία μεταξύ των σκιωδών για την ε, οδηγία για την ε, ανάκαμψη και εξυγίανση. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή και χωρίς να καλύψω το χρόνο που μου έχετε δοθεί να ευχαριστήσω τους σκιώδεις γιατί έκαναν πολύ καλή δουλειά και συνέβαλαν σημαντικά για το σημερινό θέμα, πρόεδρε. Δύο ερωτήσει θέλω να θέσω στους προσκεκριμένους μας. Πρώτον, τι μάθαμε, τι μαθαίνουμε από αυτό που έγινε στην Κύπρο. Ένα, για το πώς συζητούμε τα θέματα της στήρησης ή της αναβολής εφαρμογής των κανόνων του, Συμφώνου Σταθερότητας. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και σε κάποια αυτό που τελικά το έχουμε στερεότυπο, κάνουμε στερεότυπο λιτότητα ανάπτυξη ή ανάπτυξη και ε, τήρηση των κανόνων. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά αν υπάρχει προσδοκία επίτευξη των αποτελεσμάτων αλλά και αν πρέπει να αναλυφθεί άμεση δράση. Και αυτό που βλέπουμε για την Κύπρο είναι το τι συμβαίνει όταν δεν αναλαμβάνεται δράση και αν δεν τηρούνται οι κανόνες. Και τα αποτελέσματα είναι όπως βλέπουμε τραγικά με σοβαρές επιπτώσεις για μια χώρα. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο προσκεκλημένους μας τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε ως πως το πώς η, Επιτροπή, πώς η Επιτροπή θα απαιτεί από τα κράτη να τηρούν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Και σε σένα και σε εσάς κύριε Επίτροπε να ρωτήσω, όταν η Επιτροπή αναβάλει την τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, την υλοποίηση μάλλον των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας σε κάποια κράτη, είστε βέβαιοι ότι τώρα, απόλυτα βέβαιοι ότι τώρα να λαμβάνουν τις δράσεις που είναι αναγκαίες για να δικαιολογήσετε αυτή την καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Πρώτον, να σας συγχαρώ και σας και τους κοιόδης εισηγητές στην Επιτροπή σας για τα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις και να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, διότι η οδηγία αυτή είναι πράγματι ένα κρίσιμο στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης που χτίζουμε αυτή τη στιγμή για το ερώτημά σας ως προς τα διδάγματα που μάθαμε για την δημοσιονομική μας πολιτική. Συμφωνώ ότι τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ότι δίνουμε έμφαση σε μια μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και σε διαθωτική αξιολόγηση των δημοσίων οικονομικών όχι μόνο σε τήρηση των ονομαστικών στόχων, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό και ουσιώδες τα κράτη-μέλη να εξασφαλίζουν ότι όταν υπάρχει βραδύτερη δημοσιονομική προσαρμογή να είναι μια πολιτική αξιόπιστη. Η τροποποίηση πολιτικών έχει καταστεί δυνατή για δύο-τρεις λόγους. Πρώτον, διότι στην Ευρώπη τα κράτη-μέλη έχουν αυξημένη αξιοπιστία στην δημοσιονομική της, ε, δημοσιονομική τους πολιτική και επιτρέπει να λάβουν αποφάσεις υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεύτερον, λόγω της αποφασιστικής δράσης που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να σταθεροποιήσει την αγορά, τις αγορές και τρίτον, διότι υπάρχει ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση που μας παρέχει ένα πιο ανθεκτικό μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προσαρμογής των δημοσιονομικών πολιτικών και πρόθεσης των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Κατά την άποψή μου, η αύξηση, η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και όλο το εργαλείο, το κουτί εργαλειών που έχουμε στη διάθεσή μας παρέχουν επαρκή ε, επαρκής δυνατότητας για να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Εμείς θα παρουσιάσουμε την αξιολόγηση μας για τα, την πραγματική υλοποιηθήσα δράση στο τέλος του μήνα, μαζί με προστάσει για διαφορετικέ μεταρρυθμίσει και δημοσιονομικέ πολιτικές. Και περιμένω με χαρά να επανέλθω στην Επιτροπή σα, Έχουμε βάλει μια ημερομηνία αρχέ Ιουνίου νομίζω για να, συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τι συζητήσει αυτέ. Επίτροπε. Είστε απόλυτα βέβαιο ότι τα κράτη-μέλη που αναβάλουν, παίρνουν τις αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στην, στην αναβολή. Κοιτάξτε, εν γέννη, τίποτα ποτέ δεν είναι απολύτως εξασφαλισμένο. Όσον αφορά τώρα τα κράτη-μέλη, για τα οποία έχουμε προτείνει μία παράταση της περίοδου διόρθωσης των υπερβολικών ελλημάτων, για τα κράτη αυτά μέλη περιμένουμε ότι θα χρησιμοποιήσουν το χρόνο αυτός μια νέα ευκαιρία για να κάνουν τις απαραίτητες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Σε πολλές χώρες είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν πολύ θαραλέες αποφάσεις προκειμένου να δοθεί νέα όθηση στην οικονομική ανάκαμψη, καθώς επίσης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόμαστε σήμερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε αν γίνονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και αν εκτελούνται στο ίδιο πλαίσιο και απαραίτητες δημοσιονομικές προσαρμογές. Θα σας έλεγα για παράδειγμα όσον αφορά τη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η χώρα αυτή όντως να προχωρήσει σε πιστικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να καταφέρει να αυξήσει την οικονομική της ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πρόεδρος, συγγνώμη, ήδη δαπανίσατε 7 λεπτά ενώ είχατε 5 μόνο και πρέπει να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να μιλήσει και ο Πάμπλο και πρέπει να ολοκληρωθεί και η συνεδρίασή μας στις 11 και 4. Αν κάνατε πολύπλοκες ερωτήσεις, καταλαβαίνετε ότι και οι απαντήσεις καταλαμβάνουν περισσότερο χρόνο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να απαντήσει σε ερωτήσει που ήδη ακούστηκαν. Ας διαδικαστικό τότε, να σας επενθυμίσω ότι μιλάμε σήμερα εδώ πέρα για την Τρόικα και το όλο χρονοδιάγραμμα που έχει να κάνει με το σύμφωνο σταθερότητας για τη Γαλλία δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο συζήτηση τη Τρόικα. Χαίρομαι για την απάντηση του κυρίου Ρεν, αλλά πάντω δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η ερώτηση αυτή και η απάντηση αυτή ακούστηκε σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση. Πρόεδρο, ε, κοιτάξτε, προσπάθησα να σπιθαρχήσω λίγο, ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ο κύριος Γκοζές, ζητώ συγγνώμη, μιλήσαμε για τα διδάγματα της κρίσης. Έχουμε κάθε δικαίωμα να θέτουμε ερωτήσεις για τα διδάγματα που αντλούμε από την κρίση. Με την άδειά σας, κυρία Πρόεδρε, θέλω σύντομα να απαντήσω στην ερώτησή σας. Κατά την άποψή μας, και αυτό σχετίζεται και με, τα προγράμμα, με τις χώρες που εντάσσονται σε πρόγραμμα στήριξης και σε αυτές που δεν εντάσσονται σε πρόγραμμα στήριξης, δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κατονομάσουμε και να καταδείξουμε καμία χώρα. Θεωρούμε ότι η όλη συζήτηση που γίνεται για τη λιτότητα δεν είναι σωστή, γιατί δεν θα πρέπει να τασόμαστε υπέρ και κατά. Κανείς δεν έχει δίκιο ή άδικο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη σε μια γυράσκουσα κοινωνία. Κατά την άποψή μας λοιπόν, χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική πολιτική που ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες σταθερότητας του ενιαίου νομίσματος. Και αυτή η στάση μας δεν έχει τροποποιηθεί καθόλου από τις εξελίξεις στην Κύπρο σε κάποια άλλη χώρα. Μάλιστα έχει ενδυναμωθεί η στάση μας αυτή. Γιατί από τη μια προσπαθούμε να έχουμε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη και όλοι το ανέφερε αυτό. Από την άλλη, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι ένα γεγονός το οποίο πλέον πρέπει να αποδεχθούμε και θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια σε πολλές χώρες, γιατί έχουμε πάρα πολλές χώρες με πολύ μεγάλο χρέος. Μόνο πέντε είναι οι χώρες οι οποίες έχουν χρέος κάτω του 6%, κάτω από το κατόφλι του 6%. Η Σλοβενία, η Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Εσθονία. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε πολλές άλλες χώρες δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα κρατών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μία υγιή δημοσιονομική πολιτική. Υπάρχει ένα κατόφλι το οποίο θέτουν ε, όχι εμείς ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι ίδιες οι αγορές. και έχουμε το δύσκολο καθήκον, όλοι και οι συνάδελφοί του, να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπεται στα πλαίσια του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, χωρίς όμως να χάνουμε την προοπτική του να φτάσουμε στο 60% χρέος δηλαδή ως προς το ΑΕΠ. Και αυτό έχει εγκρίνει και η κοινοτική νομοθεσία η οποία έχει οθετηθεί εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος ο κύριος Σάντσες Περέδο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Εν όψη του μέλλοντος περισσότερο θέλω να μιλήσω για την βιωσιμότητα των προγραμμάτων βοήθειας και τους όρους για να πετύχουν. Το Δέλτα Νιτάφη είπε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη είναι το οικονομικό κλίμα. Από το ξεκίνημα της κρίσης οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν όχι μόνο μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερε θέσει εργασία, αλλά και μια θετική εξέλιξη του συνολικού χρέου του. Αυξήθηκε περισσότερο το δημόσιο χρέο, αλλά μειώθηκε το ιδιωτικό χρέο, κάτι που δεν πετύχαμε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, θα προσανατολιστεί η μακροοικονομική πολιτική για να αναπροσανατολιστεί για να υπάρχει επιτυχία. Δεύτερον, επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις για να απτυχθούν θέλουν πιστώσεις, άρα χρηματοδότηση, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται πάρα πολύ από τραπεζική χρηματοδότηση. Θα γίνει κάτι ούτω ώστε οι χώρε που υφίστανται αυτή την χρηματοοικονομική βοήθεια να έχουν πραγματική χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. Τρίτον, οικογένειε. Αποφεύθηκε να δεν συζητήθηκε ε, η ζημιά που η πέστησαν οι οικογένειες των μικροκατατεθών και στη ρευστότητά τους. Αλλά πάμε, ας πάμε και παραπέρα. Υπάρχει η οικονομική βοήθεια πρέπει να φτάσει τόσο ώστε να εξασφαλίσει την ε, βιωσιμότητα και τη φαραγγιότητα των οικογενειών, ιδίω των πλέον ευάλωτων. Αυτές είναι τις ερωτήσεις μου. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. τις εντάσσεω στην κατηγορία τι διδάγματα αντλούμε από την κατάσταση στην Κύπρο και τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Θέτεται ένα σημαντικότατο θέμα. την χρηματοοικονομική παγίδα ή τους υπερβολικά αυστηρούς κανόνες που υφίστανται πολλές περιοχές αυτή τη στιγμή. Η οικονομική ιστορία, κατά την άποψή μου, δεν αναγνωρίζει καταστάσεις όπου επιτρέπεται, μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη χωρίς πιστοτική ανάπτυξη. Στην Ευρώπη παρόμοιες επιχειρήσεις ή παρόμοιες οικογένειες αλλά κυρίως επιχειρήσεις παίρνουν δάνεια που οι όροι των οποίων είναι πολύ ψηλότεροι στη Νότια Ευρώπη από ό,τι αλλού. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό κάθε χρηματοοικονομικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να προσπαθεί στο πλαίσιο της, ε, των αρμοδιοτήτων τους να αντιμετωπίσει την ε, παγίδα ρευστότητα, ιδίω για την Νότια Ευρώπη. Μιλήσατε επίσης, συγκρίνετε μάλλον την Ευρώπη με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν δύο διαφορέ για την διαχείριση τη κρίσεω και την οικονομική ανάπτυξη. Στη ΣΥΠΑ οι ΙΠΑ μπήκαν στην κρίση νωρίτερα. Το 2007 τους έπληξε η οικονομική κρίση και το 8 ακόμα βαθύτερα. Στην Ένωση η κρίση ήρθε το 2009 ως χρηματοοικονομική και το 2010 ως κρίση χρέους πραγματικά. Δεύτερη διαφορά. Στη ΣΥΠΑ, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε προς όφελός τους, στη ΣΥΠΑ ολοκλήρωσαν την οικονομική επισκευή τους γρήγορα και αποτελεσματικά με ε, μεγάλο μπαζούκα όταν έκλεισε η Lehman Brothers το 2008. Η οικονομική αυτή ε, επισκευή έγινε κατά βάση το 2009 που επέτρεψε καλύτερες συνθήκες για την απασχόληση και την ανάκαμψη το μάθημα για μας είναι ότι η οικονομική επισκευή, η χρηματοοικονομική επισκευή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και ανακεφαλαίωση του τραπεζικού τομέα, να δημιουργήσουμε μια τραπεζική ένωση και να λύσουμε την παγίδα ρευστότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Νότια Ευρώπη. Μπορείτε κι εσείς να απαντήσετε κύριε Σμούσεν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δύο θέματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τον δανεισμό όλοι θα επαναλάβω αυτά που είπα όλοι στο τέλος όταν σε έκανε τη σύγκριση με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ήταν ταχύτερε στην εκαθάριση των τραπεζικών ισολογισμών και στην ακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη τρενάρει έως ότου υπάρχει, υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ισολογισμούς των τραπεζών δεν θα υπάρξει δανεισμός στα επίπεδα που ξέραμε πριν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταστήσουμε, που το καθιστούμε σαφές στο νομοθετικό κείμενο για την τραπεζική εποπτεία πρέπει αυτό να γίνει πριν ξεκινήσει ο ενιαίο χρηματοοικονομικός ε, μηχανισμός εποπτείας και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για την εκαθάριση των τραπεζικών ισολογισμών στην Ευρώπη. Για την, παροχή, για την πιστοτική παροχή, ιδίω προ τι μικρομεσαίες επιχείρησει. Προφανώ σε κάποια μέρη της Ευρωζώνης, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα. Εμείς στην τράπεζα προσπαθήσαμε να δούμε με ανοιχτό πνεύμα τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Σχετίζεται με την παροχή ρευστότητα στις τράπεζες, κάναμε αρκετά εδώ και κατά μέσο όρο, ωστόσο και αυτό είναι ένα πρόβλημα, φαίνεται ότι η ρευστότητα δεν εμποδίζει τον τραπεζικό αδενανισμό. Το θέμα είναι είτε ε, αύξηση είτε έλλειψη κεφαλαίου είτε φόβος του κινδύνου. Αυτό ε, είναι που εμποδίζει τον, βασικά τον δανεισμό, που δεν είναι δική δική μας δουλειά. Ίσως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορεί να βοηθήσει. Πάντως μέσα στο πλαίσιο του δικού μας, ε, της δικής μας εντολής θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά θέσετε ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα βασικό ζήτημα για πολλές χώρες. Η κυρία Κράτσε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θεσμικά όργανα και η ερώτησή μου σχετίζεται και με αυτά που μόλις είπαμε για το θέμα της ρευστότητας και της ικανότητας των τραπεζών να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία. Προς το παρόν βλέπουμε ότι θίγονται από την ευρωπαϊκή οικονομία και την ύφεση και φυσικά συνδέεται η ερώτησή μου και με την προβλεψιμότητα που είδαμε ότι μας έλειψε και στην περίπτωση της Κύπρου, να μην επανέλθω στις αδυναμίες που ήδη ε, τονίστηκαν όπως ανεδείχθηκαν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις σχέσεις των τραπεζών στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη Βασιλεία 3. Μου έκανε εντύπωση μια πρόσφατη μελέτη της HBC η οποία λέει ότι ε, εκτιμάει ότι 3,33 ευρώ θα είναι το κεφάλαιο που θα πρέπει να βρεθεί όχι υπό τη μορφή μετοχών από την αγορά για να απορροφηθούν οι ζημιές σε περίπτωση διάσωσης εσωτερικής προέλευσης. Ήθελα να ρωτήσω καταρχάς αν έχετε δικές σας εκτιμήσεις ή πώς ε, ε, εκτιμάτε αυτά τα, τα στοιχεία και δεύτερον, εάν θεωρείτε την, ότι οι τράπεζές μας έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε απαιτήσει τη Βασιλεία 3 και επίση, αν ε, η πιθανή κλιμάκωση επισφαλιών στην οποία ήδη ε, αναφερθήκατε ότι επιβαρύνει τι τράπεζε, θα μπορούσε να έχει επιπτώσει στην εξασφάλιση των απαιτούμενων ε, κεφαλαίων και τι ιδιαίτερε προσπάθειε που πρέπει να κάνουν οι τράπεζε, άρα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στι ανάγκε τη αγορά. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε, κυρία Κράτσα. Κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι οι περισσότερες ερωτήσεις είναι για τον κύριο Άσμουσεν που θα απαντήσει μετά εγώ θα απαντήσω σε αυτό που είπατε για την ανάγκη εξασφάλισης ρευστότητας για την πραγματική οικονομία. Και με αυτή την ευκαιρία υπογραμμίζω τη σημασία της αναδιάρθρωσης και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στο ελληνικό πρόγραμμα. Γιατί αυτό είναι ουσιώδες να έχουμε δηλαδή ε, ροή πιστώσεων και να υπάρξει δανειοδότηση απαιτούμενη ε, από την οικονομία και για την ανάπτυξη. Ε, βεβαίως εδώ υπάρχει και σύνδεση μεγάλη με την Κύπρο, γιατί τα ελληνικά υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών, των τριών, επολύθησαν διότι η πώληση συνέβαλε κατά πολύ στη μείωση του μεγέθους ε, των τραπεζών στην Κύπρο και να σταματήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης ε, της κρίσης ε, από τη μια χώρα στην άλλη. Δεύτερον, δεδομένη της συνολική κατάστασης στην Κύπρο υπήρχε ο φόβος ότι οι Έλληνες καταθέτες θα μπορούσαν να, πάνε, να πάρουν τα χρήματά τους και να τα πάνε αλλού και οι κυπριακές τράπεζες και έτσι η πώληση των ε, ελληνικών υποκαταστημάτων μπορεί να ήταν δαπανηρή, αλλά ήταν λιγότερο δαπανηρή από τη διατήρηση των υποκαταστημάτων που θα μπορούσαν να καταρρεύσουν με, λόγω μαζικών ε, ε, αναλήψεων, bank run. Επίσης οι δυσκολίες των ελληνικών ε, υποκαταστημάτων θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την εμπιστοσύνη στον ελληνικό τραπεζικό τομέα που τώρα μετά από δύο χρόνια μεγάλης καθοδικής τάσης τώρα ανακτά ε, έναν αριθμό καταθετών που είναι σημαντικό αυτό για το, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Η Τρόικα εμεθάρρυνε και την ελληνική και την κυπριακή πλευρά να διαπραγματευτούν επί της πωλήσεως αυτών των υποκαταστημάτων. Έγιναν διμερείς διαπραγματεύσεις και η Τρόικα έδρασε διευκολυντικά διαμεσολαβητικά και στις 26 Μαρτίου νομίζω ελήφθη σχετική απόφαση για την πώληση. Ε, ευχαριστώ επιτροπε ο κύριος Σάσμουσεν. Ευχαριστώ. Κυρία Κράτσα, σχετικά με την πρώτη σας ερώτηση δεν ξέρω ακριβώς σε ποια μελέτη αναφέρεστε που είπατε τα 3,5 δις. Καλό είναι να το διευκρινίσουμε αυτό και να απαντήσω μετά την ακρόαση. Ε, κάποια στιγμή σε, μετέπειτα χρόνο. Τώρα, γενικότερα, για το Tier 3. Είμαστε επεπισμένοι ότι βρίσκεται στο, στην καρδιά του προβλήματος της, και της ατζέντα της μεταρρύθμισης και έχει να κάνει με την ε, ε, εξυγίανση των ισολογισμών της τράπεζας, η βασιλιατρία, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν εγγυάται την καλύτερη ποιότητα και ποσότητα κεφαλαίων ε, στις τράπεζες. Και αν κατάλαβα καλά, ε, ε, ερωτάτε εάν απαιτούμε υπερβολικά πολλά πράγματα από τις τράπεζες. Υπάρχουν στοιχεία μετά, από το τέλος του 2008 και μέχρι τέλος ότι κατά μέσον όρο η κεφαλαιακή κατάσταση με βάση το Tier 1 και το βασικό δίκτυο ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών αυξήθηκε πολύ αλλά αυτό που βλέπουμε παράλληλα είναι ότι ε, τα κεφαλαϊκά αποθέματα ε, είναι άνισα κατανεμημένα μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών και αυτό θέτει κάποια ερωτήματα από τους επενδυτές και μπορεί να εμποδίσει την επανεκκίνηση ε, του δανεισμού. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προσεκτική ισορροπία και μου φαίνεται ότι αυτό επετεύχθη. Οι υψηλότερε κεφαλαιακές ανάγκε που απαιτούνται για ε, την ε, σταθερότητα και από την άλλη πλευρά η παροχή δανείων που είναι βασικό καθήκον ε, των τραπεζών προς την οικονομία. Η Βασιλεία τρία με τις τελευταίες τροποποιήσεις που είδα για την κεφαλαιακή επάρκεια, για το δανεισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπόρεσε να, επαν... να, να ξαναβρει ε, την ισορροπία που είχε χαθεί. Θα σας απαντήσω στην άλλη ερώτηση ε, αργότερα. Ε, ο κύριος Σάιμον και εγώ να κάνουμε τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν ε, και οι δύο μαζί. Ο κύριος Σάιμον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Ασμούσεν. Ε, μιλάμε για την Τραπεζική Ένωση ε, που την θεωρείται επιθυμητή. Αυτό το οποίο με κάνει να διστάζω λίγο ως εισηγητής για την εξασφάλιση των καταθέσεων ε, είναι ότι αναδείξατε τη σημασία της εποπτείας και της νομοθεσίας για την εξυγίανση. Η, Τραπεζική Ένωση αποτελείται από τρία μέρη και από την εγγύηση των καταθέσεων. Ε, δεν θα μιλήσω εδώ για τα ταμεία ε, εγγύηση των καταθέσεων, αλλά για την πρόταση ε, νομοθεσίας που κάνει σχετικά η Κομισιόν. Και το, το ύψος των ταμείων, των κεφαλαίων, ε, που θα χρειαστούν ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ δεν υπάρχουν διστάμενες απόψεις, ε, έχουμε ε, σύμπτωση απόψεων και το Κοινοβούλιο τροποποίησε σε πρώτη ανάγνωση την, πρώτη, πρόταση της Κομισιόν και την ψήφισε με 85% όμως μπλοκαρίστηκε η διαδικασία στο Συμβούλιο μεταξύ άλλων για το πόσο στα σταέρεο θα πρέπει να είναι ε, ένα τέτοιο ταμείο και πόσο γρήγορα πρέπει να συσταθεί. Νομίζω ότι αν παρουσιάσει εδώ η Τρόικα τις προοπτικές για το μέλλον θα θέλαμε να μας πούν δυο ξεκάθαρα ε, λόγια για το Συμβούλιο και τη διαδικασία ε, λήψης απόφασης για το Ταμείο, το ύψος των κονδυλίων που θα διαθέτει, και να μας πει και πόσο γρήγορα ε, θα ε, αποκατασταθεί η επιθυμητή σταθερότητα. Ευχαριστώ κύριε Σαϊόνμον. Η ερώτησή μου είναι προς τον κύριο Σμούσεν. Συμφωνώ μαζί σας ε, και με τον Επίτροπο για την ανάγκη να υπάρξει ενιαίος επόπτης και μηχανισμός εξυγίανσης καθώς και την σημασία της δημοσιονομικής εξυγένσης και των μεταρρυθμίσεων. Ενώ ωστόσο οι χρηματοοικονομικές αγορές συνεχίζουν να είναι κατακαιρματισμένες, δεν θα χρησιμεύσει πάρα πολύ όλα αυτά για να φτάσει η τραπεζική πίστη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις οικογένειες. Μιλούσατε για εμπιστοσύνη κύριε Σμούσεν, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο ακριβώς βλάπτει την εμπιστοσύνη και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την αποκατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Ε, η μείωση των επιτοκίων είναι καλό μήνυμα, καλό νέο. Έχω αμφιβολίες ωστόσο αν αυτό θα έχει επιπτώσει στην πραγματική οικονομία δεδομένων των, δεδομένης του καρματισμού της αγοράς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο ακόμα περαιτέρω ε, οξύνει και δυσχεραίνει την, τον κατακαιρματισμό των αγορών. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε στην τράπεζα κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να πάψουν να είναι οι αγορές ε, κατακαιρματισμένες, ιδιαίτερα ό,τι αφορά την ε, πίστοση προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα και κάποια σχόλιά σας για κάποιες πληροφορίες που είδα στον γερμανικό τύπο σήμερα που λέει στα αγγλικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσβλέπει στην εξαγορά κακών δανείων από νοτιοευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα ο Επίτροπος και μετά ο κύριος Ασμούσεν. Ευχαριστώ. Thank you. Think... Uh, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δύο από τις ερωτήσεις σας αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φαντάζομαι ότι ο Γιώργος θα απαντήσει σε αυτές. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Σάιμον, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας πραγματικά. Πρέπει να προχωρήσουμε με την όλη έννοια της Τραπεζικής Ένωσης, να ολοκληρώσουμε το μηχανισμό αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν ως προς το στόχο αυτό και νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπαρνιέ, ο συνάδελφός μου, επεξεργάζεται έναν κοινό μηχανισμό εξυγίανσης και θα παρουσιάσουμε πριν το καλοκαίρι μια νομοθετική πρόταση για το ζήτημα αυτό. Και λίγο αργότερα, μετά από ενδελεχή προετοιμασία, θα υποβάλουμε μια πρόταση για ένα κοινό ταμείο εγγύησης των καταθέσεων. Αυτό όμως θα μας απασχολήσει στο απότερο μέλλον και όχι άμεσα και αποτελεί πάντως πολύ σημαντικό στοιχείο του οικοδομήματος της Τραπεζικής Ένωσης. Ένα άλλο μάθημα το οποίο μπορούμε να μάθουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν το 1934 στη χώρα αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντικές προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καταθέσεις και να αποφευχθεί κάποια περαιτέρω τραπεζική κρίση και επίσης οχυρώθηκε καλύτερα η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της χώρας η οποία δεν ιδιωτεί προς τις υπόλοιπες τράπεζες. Πρέπει να σας πω ότι ε, οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν ε, να κάνουν με την αρμοδιότητα του κυρίου Άσμουσεν, καθότι πρόκειται τώρα για την τελευταία μου παρέμβαση. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, αυτή την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, και θα ήθελα πραγματικά να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον και ας προσπαθήσουμε από κοινού να μελετήσουμε καλύτερα τα διδάγματα της πρόσφατης αυτής εμπειρίας και να καταλήξουμε σε κάποια θετικά συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριε αν έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ως προς το ερώτημα του κυρίου Σάιμον. Γνωρίζω την ενεξελίξη συζήτηση για την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι επιτάπητος εδώ και κάποιο καιρό βέβαια. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις στο Συμβούλιο, έχω παρακολουθήσει πολλέ συζητήσει στο Συμβούλιο. Η δική μα η πλευρά υποστηρίζει πάντα το στοιχείο αυτό που έχει να κάνει με το κοινό Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων. Θέλουμε το κοινό αυτό Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων να γίνει πραγματικότητα και ο κύριος ε, Όλι αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό ταμείο των καταθέσεων στο απότερο μέλλον ως αναπόσπαστο τμήμα της α, Τραπεζικής Ένωσης. Προκειμένου να έχουμε μια Τραπεζική Ένωση χρειαζόμαστε ε, να κλείσουμε επιτυχία όλα τα επιμέρους στοιχεία της. Προφανώς θα πρέπει να κοιτάμε και τα επιμέρους στοιχεία της Τραπεζικής αυτής Ένωσης, αλλά και σφαιρικά την όλη Τραπεζική Ένωση. Ως προς ε, το ερώτημα του Προέδρου, Όντως, οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι ακόμα κατακαιρματισμένες ε, στην Ευρωζώνη και βέβαια αυτό δυσχεραίνει την ε, καλύτερη διαχείριση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα επιτόκια. Ήδη όμως από πέρυσι το καλοκαίρι βλέπουμε ότι ο κατακαιρματισμός αυτός έχει κάπως μειωθεί. Υφίσταται ακόμα, ακόμα μας ανησυχεί αλλά αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι έχουν ε, αναλυφθεί κάποιε δράσει από ορισμένα κράτη-μέλη, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίε ε, μείωσαν κατά τη τον κατακαιρματισμό αυτών των αγορών. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει σε ορισμένες χώρες και ιδίω ως προς τους ε, στόχους που θέτουν πλέον οι χώρες αυτές για τους ισολογισμούς τους που λένε πολλά για τον κατακαιρματισμό της, των αγορών, καθώς επίσης και για τη μην λειτουργία ή την δυσλειτουργία των διατραπεζικών συναλλαγών. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη τώρα από ό,τι πέρυσι τον Οκτώβριο. Κατά 20% έχει μειωθεί το φαινόμενο αυτό του κατακαιρματισμού. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στην απόλυτα φυσιολογική κατάσταση. Υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωσης. Αλλά έχουμε εντοπίσει ήδη κάποια βελτίωση που έχει λάβει η χώρα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα εμείς για τον κατακαιρματισμό των αγορών, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, αλλά τα περισσότερα πράγματα μπορούν να τα κάνουν οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Πώς μπορούν δηλαδή να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς επίσης και των καταναλωτών. Τα περισσότερα μη τυπικά μέτρα, non-standard measures, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Τρενκητή Τράπεζα, το μέσο για παράδειγμα OTN καθώς επίσης και άλλα μέσα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει δεν πρόκειται για τα συνήθι συμβατικά μας μέτρα αλλά τα χρησιμοποιήσαμε για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποιους ε, χώρους της Ευρωζώνης όπου εξαιτία του κατακαιρματισμού η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει λοιπόν μια νέα ομάδα εργαλείων που αμφισβητούνται σε κάποια μέρη της Ευρωζώνης, αλλά θεωρώ ότι είναι σωστό να έχουμε μια νομισματική πολιτική η οποία επιτέλους θα φτάνει μέχρι τα νοικοκυριά, μέχρι τις επιχειρήσεις, σε αυτό το κατακαιρματισμένο τοπίο των αγορών που έχουμε. Αν αναφερθήκατε σε ένα άρθρο που διαβάσατε σήμερα το πρωί, φαντάζομαι ότι σε ένα άρθρο της Die Welt. Κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή όλη η εργασία την οποία κάνουμε προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη δανειοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη σήμερα το πρωί το συζητήσαμε το ζήτημα αυτό θέλουμε να καταφέρουμε να καλύψουμε όλες τις δράσεις που μπορούμε να λάβουμε στα πλαίσια της εντολής μας και να έχουμε μια καλύτερη αγορά για asset-backed securities για να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη δανειοδότηση προς επιχειρήσεις αλλά με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας αυτή τη φορά, με την απαραίτητη εποπτεία. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε ακριβώς ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο προσκεκλημένους μας. Φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και ευχαριστώ τους διαδυνείς που έμειναν παραπάνω. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει στις 20 Μαΐου στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε. Τέλος της συνεδρίασης.